μπορούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Καταρχήν θέλω όλους να σας καλωσορίσω μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, μετά από την εκλογική αναμέτρηση, μετά από τις ταραγμένες πρώτες μέρες εδώ. Ελπίζω ότι να ξεκουραστήκατε και να ήρθατε με υγεία και αποφασιστικότητα για να ξαναρχίσουμε την κανονική μας εργασία στη νέα θητεία. Ξεκινάμε σήμερα τη νέα σχολική χρονιά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν όσον αφορά το σχέδιο μερίσιας διάταξη υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Όχι, δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εγκρίνεται το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Δεύτερον, έχουμε κάποια πρακτικά της 10ης Ιουλίου. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχετε τα πρακτικά αυτά στο φάκελό σας. Έχετε παρατηρήσει σχόλια. Ως συνήθως θεωρούμε λοιπόν ότι τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, αν κάτι σκεφτείτε μπορείτε να μου το υποβάλλετε. Περνάω στο σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα σας μιλήσω καταρχήν για την διερμηνία. Η διερμηνία έχουμε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, φιλανδικά, τσεχικά, ουγγρικά, λετονικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ρουμανικά. Αυτές είναι οι γλώσσες για τις οποίες έχουμε διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους διερμηνείς για την συμμετοχή τους. Επίσης θέλω να σας πω, να σας υπενθυμίσω ότι αναμεταδίδεται ζωντανά η σημερινή μας συνεδρίαση και βεβαίως θα ψηφίσουμε καταρχήν, και αυτό είναι το σημείο 4 της σημερινής της διάταξης, για τις τροπολογίες ε, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, όλα τα τμήματα Πρόκειται για τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε ξεχωριστά την κάθε τροπολογία και δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία ακριβώς επειδή πρόκειται για τροπολογίες που αφορούν τον προϋπολογισμό. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου και βεβαίως θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και τις τελικές μας θέσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό όταν ψηφίσουμε και όταν ξέρουμε ποιες είναι οι τροπολογίες αυτές που έχουν περάσει, γνωρίζουμε επίσης και όλες τις θέσεις Επιτροπής, δεν χρειάζεται σήμερα όμως η τελική εντολή να δοθεί. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Θέλει να πάρει το λόγο η συγγήτρια. Πέτρα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Στην αρχή της κάθε θητείας υπάρχει μια σχετική σύγχυση όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, την αξιολόγησή τους. Εγώ έκανα μια γενικότερη παρουσίαση αυτής της έκθεσης λέγοντας ότι δεν θα στηρίξουμε πιλωτικά προγράμματα τα οποία οδηγούν σε κατηγοριοποίηση στις κατηγορίες C και D. Και μάλιστα ε, δώσαμε και κάποιες διευκρινήσεις. Η κατηγορία C δεν σημαίνει ότι κάποιο πρόγραμμα δεν είναι αξιόλογο, είναι κακό. Σημαίνει ότι ουσιαστικά η χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων θα πρέπει να επανεξεταστεί. Σε καμία περίπτωση λοιπόν η κατηγορία C δεν αναφέρεται στην ποιότητα του εν λόγω πιλωτικού προγράμματος, αλλά σε θέμα τρόπου χρηματοδότησης. Εγώ έβαλα μείον λοιπόν σε όλες αυτές τις κατηγορίες C και D. Σας εξηγώ όμως ότι αυτό δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ποιότητα του εν λόγω πιλωτικού προγράμματος. Μπορεί σε καμία σε μια άλλη περίπτωση να το είχαμε υποστηρίξει και εγκρίνει. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Έχετε μαζί σας όλοι τις κάρτε κάρτες σας. Ναι. Ψηφίζουμε καταρχήν την τροπολογία κουλ cool 5900 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5901 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5902 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5903 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στο 5909 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το 5906 ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά αποχές εγκρίνεται. 5907 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η 59.05 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 59.10 59.04 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα το είχαμε ψηφίσει. Και τώρα περνάμε στην 5910 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5908 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5912 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 59-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59-19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59-20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59-21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ταυτόσημα με την 23 και περνάμε στην 59-22. Αποσύρθηκε όμως. 59-24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59-26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59-27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ταυτόσιμο με το 28, 59-29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59-30 59,30 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρινεται 59,31 59-31 υπέρ, κατά, αποχές 59,32 59-32, ταυτόσιμο με 33 υπέρ, κατά, αποχές 59,34 και 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 59-36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 59-51 και 52, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στην προφορική τροπολογία 59-50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59, 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59, 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59, 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5941 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5942 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5943 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα περνάμε στην 5944 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59... 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59-47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59-48 αποσύρεται, 59-45 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59-55 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59-53, ταυτόσιμη με την 54 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59-58 58. Όχι. «56 καταπίπτει, 59-58 υπέρ». Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59-60 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, καταπίπτει. Περνάμε στην 61. 59-61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-64 αποσύρθηκε και περνάμε στην 59-65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59-66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59-67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59-68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59-69 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59-70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 59-71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59-72 κατά αποχές εγκρίνεται 59-73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59-74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5975 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5976 ταυτόσημη με την 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5978 έχει αποσυρθεί. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία για σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στον ε, γενικό προϋπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το 2020, όλα τα τμήματα. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση την οποία θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Προλογισμού. Η εισηγήτρια με τους αρμόδιους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμού έχουν επεξεργαστεί το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020. Υπάρχουν τεχνικές ουσιαστικά τροπολογίες. Τα μηνύματα, τα πολιτικά είναι πολύ συγκεκριμένα που πρέπει να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ όταν βγαίνετε να είστε σιωπηλοί έτσι ώστε να μπορούμε να ακούσουμε πριν δώσω το λόγο όμως στην εισηγήτρια, θέλω να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 12 τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. Τη Δευτέρα στις 12, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου υποβολή για τις τροπολογίες προθεσμία. Η Πέτρα Κάμερφερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Σαμπίν, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι όπως ακούσατε. Έχουμε ψηφίσει τώρα πια για το σχέδιο προϋπολογισμού για τις τροπολογίες και τώρα μπορούμε λιγάκι να συζητήσουμε για την γνωμοδότησή μας, δηλαδή το πολιτικό κείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει τις ιδέες μας. Βεβαίως ε, είναι αυτονόητο ότι θα λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα των, της ψηφοφορίας, ποιες δηλαδή οι τροπολογίες πέρασαν και ποιες απεριφθήσαν. Σας είχα παρουσιάσει με σαφήνεια νομίζω στη συνάντησή μας τον Ιούλιο τις προτεραιότητές μας. Ο Γενικός Προπολογισμός όπως ε, υπευλήθη από την Επιτροπή στηρίζεται από εμάς σε αντίθεση με τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο και θεωρώ πραγματικά ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις ε, συγκεκριμένες περικοπές. Ξέρουμε όλοι τα σημαντικά προγράμματα, το Erasmus, το Erasmus Plus, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σώμα, ε, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μειωθούν τα ποσά για όλα αυτά τα πολύ συμβολικά και πολύ σημαντικά προγράμματα, όπως παραδείγματο χάρη η Δημιουργική Ευρώπη, η Ευρώπη των Πολιτών, ανδρών και γυναικών. Οι συγκεκριμένες μας προτάσεις είναι και για το Erasmus Plus να αυξηθούν τα ποσά κατά 10%. Βλέπετε ότι υπάρχει και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό θα το στηρίξουμε και στον τριμερή διάλογο. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο. Για το Erasmus ζητάμε τριπλασιασμό, για το Creative Europe ζητάμε διπλασιασμό, καθώς και το σώμα αλληλεγγύης, το οποίο θέλουμε να χρηματοδοτηθεί με ένα ποσό το οποίο θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί και όχι να συρρυκνωθεί. Βεβαίως ε, έχουμε και κάποιες πιο αυστηρές, αν θέλετε, παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα αναφέρομαι και θα το είδατε στο κείμενό μου στη χρηματοδότηση του Euronews καθώς και των ε, άλλων προγραμμάτων που αφορούν τα πολυμέσα και τις πλατφόρμες. Πιστεύω ότι και αύριο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό καθότι η στάση μας είναι αυστηρή οι επικρίσεις όχι μόνο από τη δική μας Επιτροπή αλλά και από άλλες Επιτροπές του Κοινοβουλίου νομίζω είναι εξαιρετικά αν θέλετε, αυστηρή. Υπάρχουν σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες της Ευρώπης που δεν έχουν πρόσβαση στο Euronews και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η οικονομική κατάσταση, αν θέλετε, η οποία κανονικά θα πρέπει να επιτηρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Euronews, δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ανεξαρτησία και σε καμία περίπτωση εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι τηρήθηκαν ε, τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο και όπως ακριβώς έχουν τεθεί για την ετήσια παρακολούθηση και εποπτεία. Οι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει στην ε, ε, ετήσια έκθεσή τους ότι όλο και περισσότερο αν θέλετε, χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς, από ιδιωτικούς επενδυτές. Περίπου το 58% των, ε, της χρηματοδότησης προέρχεται από τέτοιους πόρους. Αυτό δεν είναι καθόλου ε, ευχάριστο. Βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Βεβαίως, ε, και αυτό θα είναι και το τελικό μου συμπέρασμα, λίγα άλλαξαν, λίγο ελήφθησαν υπόψη οι δικές μας παρατηρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει από τη στιγμή που δεν ακούγονται οι δικές μας παρατηρήσεις, από τη στιγμή που δεν μας λαμβάνουν υπόψη, να σταματήσουμε αυτήν την συνεργασία με το Euronews. Από τη στιγμή που δεν αντικατοπτρίζεται πλέον, αν θέλετε, μια οπτική γωνία την οποία θέλουμε. Ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα μια αύξηση της χρηματοδότησης τάξης του 5%, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό και με πιο σωστό τρόπο τα ποσά αυτά. Πιστεύω ότι αυτά τα εκατομμύρια που κάθε χρόνο πηγαίνουν προς το γύρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να εκπληρώσουν το σκοπό μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι ακριβώς επειδή ο στόχος μας είναι οι νέοι, είναι η κοινωνία της Ευρώπης ε, να αποκτήσει περισσότερη δημιουργικότητα, είναι ο αθλητισμός, είναι η στήριξη όλων αυτών των τομέων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, Πέτρα. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στους κοιόδες εισηγητές. Κρίστιαν, έλα, δεν είναι εδώ. Η κυρία Σόντροβα θα τον αντικαταστήσει. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Συμφωνώ απολύτως με, τον, ε, με την εισηγήτρια. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μείωση της στήριξης απαραίτητων για εμάς προγραμμάτων. Τα επιχειρήματα που προβάλλει η Επιτροπή Πολιτισμού τονίζουν την ανάγκη για επενδύσεις, την ανάγκη να επενδύσουμε στη νέα γενιά, να ενισχύσουμε το δημιουργικό πνεύμα, τους νέους δημιουργούς. Πρόκειται για προγράμματα που μας επιτρέπουν να επενδύσουμε στη νεολαία, στη νέα γενιά. Έτσι ώστε να καταλάβουν οι νέοι ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να τους προσφέρει. Τώρα για το Euronews. Να το δούμε το θέμα και μάλιστα ενδελεχώς. Να το μελετήσουμε σε βάθος. Είναι ένα κανάλι που αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τότε πρέπει πράγματι να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με αυτό. Για να μπορέσουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν εμπιστοσύνη, να μπορούν να έχουν απαραίτητες και αντικειμενικές πληροφορίες. Άρα, να εξετάσουμε ενδελεχώς και επισταμένως το θέμα της χρηματοδότησης του Euronews. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, στηρίζουμε την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λόγω, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αξιότιμη κυρία εισηγήτρια για την δουλειά Στη δική μας ομάδα στηρίζουμε την προσέγγιση της εισηγήτριας σε ό,τι έχει να κάνει με την ετούμενη αύξηση κατά 10% της επιχορήγησης για τα προγράμματα Erasmus+. Plus. για τα προγράμματα Creative Europe και Ευρώπη των πολιτών, οι περικοπές που ζητά το Συμβούλιο είναι ανησυχητικές και υπονομεύουν τον τομέα του πολιτισμού, τον τομέα της ε, δημιουργίας, αλλά υπονομεύουν και την ενότητα των Ευρωπαίων. Άλλωστε η Ευρώπη των πολιτών και το Erasmus πλάσε, γι' αυτό έγιναν και γι' αυτό σχεδιάστηκαν για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, Εμεί συμμεριζόμαστε με την άποψη αυτή για την ενίσχυση του προπολογισμού των προγραμμάτων. Με ικανοποίηση βλέπω να έχει διατυπωθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική απαραίτητη για την πρόθεση και τη διάσωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού με οριζόντα το 2020 και, στο, ε, και με βάση το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως, η χθεσινή συνάντηση των εισηγητών για τις τροπολογίες έδειξε ότι έχουμε κάποιες αποκλίνουσες απόψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη γραμμή δράσης για τα πολυμέσα. 5% αύξηση προϋπολογισμού ζητάμε για αυτή την γραμμή του, προ... προϋπολογισμού. Για τα ραδιοφωνικά δίκτυα Euronet. Ελπίζω να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμβιβαστική λύση για την κατάσταση του καναλιού Euronews που ε, απορροφά τα 3 τέταρτα της χρηματοδότησης αυτής της δράσης λείπουν τα κονδύλια, λείπει μάλλον η παρακολούθηση για το τι γίνονται τα κονδύλια που δίδονται στο Euronews από πλευράς κομισιών. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυστηρότερη πλαισίωση. Σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης που θα μιλούν για την ευρωπαϊκή ε, πραγματικότητα. Με βάση τα πρότυπά μας η εταιρική σχέση είναι ατελής και πρέπει να έχουμε εναλλακτική λύση και ένα αξιόπιστο μέσο το οποίο να είναι αντικειμενικό, να λειτουργεί με διαφάνεια και να είναι ευρωπαϊκό. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και με το ελεκτικό συνέδριο να συνεργαστούμε και να χυθεί φως σε όλη αυτή την υπόθεση. Περιμένουμε μεγάλη αγωνία και ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση, αλλά και τις απόψεις από αυτού του συναδέλφου εισηγήτριας. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια, αλλά και την πρόεδρο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κυρία Κάμερβερτ. Κάνατε εξαιρετική δουλειά διαπραγματεύεστε τον προϋπολογισμό με εμάς. Νομίζω το, το βασικό θέμα το οποίο έθιξαν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι η κατάσταση με το Euronews. Χθες συζητήσαμε ε, με λεπτομέρειες πώς να προχωρήσουμε. Όταν συντάχθηκε το πρώτο προσχέδιο, είδαμε τότε και είπαμε εκεί ότι δεν χρειάζονται χρήματα για το Euronews ή δεν υπάρχει επιθυμία να δοθούν χρήματα για το Euronews και αυτό είναι ανησυχητικό σε σύγκριση και με το τι γίνεται με το Euronet. Άρα πρέπει να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση. Θέλουμε να στηρίξουμε το Euronet, θέλουμε να ε, στηρίξουμε το ιδανικό του Euronews, δηλαδή την ε, υποκείμενη ιδέα πίσω από αυτό, δηλαδή ένα ε, κανάλι το οποίο θα αναφέρεται στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Στηρίζουμε αυτή την ιδέα βεβαίως για να μαθαίνει ο πολίτης τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά δεν μας αρέσει η ιδέα αυτό, αυτή την διοκτησία αυτού του καναλιού να την έχουν ιδιώτες επενδυτές και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Και πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα, να διορθωθεί και μάλιστα τάχιστα. Υπάρχει και το θέμα της έκθεσης για του προπολογισμού, δηλαδή πώς θα αλλάξουμε το Euronews και νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στραφεί η Επιτροπή μας στο μέλλον έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο Euronews από ό,τι έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι η συμβαστική λύση είναι καλή, να στηρίξουμε το Euronet, αλλά το πρόβλημα είναι ότι περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για συμβιβασμό. Και ε, συνεχίζουμε να δίνουμε χρήματα στο Euronews και κάποιοι από εμά δεν θέλουμε να συνεχίζει να συμβαίνει αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει πραγματικά να απασχολήσει την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αύριο έχουμε ακρόαση για το θέμα αυτό, όπως ξέρετε. Οπότε νομίζω θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το θέμα του Euronews και των επενδυτών και πώς κατανέμονται εξάλλου τα κονδύλια. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα και πιλωτικά και θα δούμε πώς και τι μπορούμε να στηρίξουμε. Αύριο νομίζω θα μπούμε εις βάθος σε αυτό το θέμα. Είναι περίπλοκο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Η Κριστίν Άντερσον έχει το λόγο. Νομίζω ότι η δική μας ομάδα μπορεί ουσιαστικά να πει ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά για να, χρησιμο... για να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους ε, οπτικοακουστικά μέσα. Νομίζω ότι από εχτες ε, που ξανασυζητήσαμε το θέμα αυτό σε μια άλλη επιτροπή είχα πει ότι, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι εδώ δεν θέλω να χαρακτηριστούμε σαν ευρωφοβικοί. Δεν θεωρώ ότι τα μέσα, τα οπτικοακουστικά μέσα είναι δημόσιο αγαθό, ότι είναι σε αυτή την περίπτωση εδώ κρατικά και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διαδίδεται μια δημόσια ή γενική άποψη χρησιμοποιώντας ε, δημόσια κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Chair. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του ECR να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την επικοδομητική της εργασία και την οργάνωση των συζητήσεων για το θέμα αυτό. Γενικά, στηρίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που δείχνει την ε, ε, γνώμη γενικά του σώματος. Μεταξύ άλλων όμως, το Έρασμος είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα της Ένωσης και χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο αυτό προκειμένου να επιτελέσει το έργο του. Κατά τον ίδιο τρόπο, συμφωνώ ότι τα κονδύλια για την Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να αποκατασταθούν στα αρχικά τους επίπεδα. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία που μόλις έγινε, η ομάδα μας είναι υπέρ της διατήρησης των απαραίτητων πόρων για τις ε, δράσεις πολυμέσων. Όμως έχουμε μία επιφύλαξη όσον αφορά τις επιδόσεις του Euronews και τις ε, σχετικές ελλείψεις εκεί. Το ελεγκτικό, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, είπε ότι υπάρχουν προβλήματα και συμφωνούμε με τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να βρούμε μια μακροπρόθεσμη λύση ούτως ώστε να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ταυτόχρονα Χαίρομαι διότι έχουν γίνει πολύ καλές προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα και προπερασκευαστικές δράσεις, κυρίως όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως όσον αφορά την ιδιοκτησία, την παιδεία, εξοικείωση με τα μέσα. Η έκθεση όμως έχει και κάποια μικρά ελαττώματα. Ε, έχουμε λοιπόν καταθέσει τροπολογίες αλλά και πάλι γενικά είναι μια πολύ καλή γνωμοδότηση και πάλι συγχαρητήρια για το επικοδομητικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, και έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι βεβαίως η παιδεία και ο πολιτισμός. Νομίζω ότι γενικά έχουμε την τάση να υποτιμούμε τη σημασία του όσον αφορά την χρηματοδότηση. Και βεβαίως και εγώ ζητάω, λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες να τους στηρίζουμε όσον αφορά την ανάπτυξη του πολιτισμού για να μπορέσουν να ε, συνειδητοποιήσουν καλύτερα την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χτες όσον αφορά το Euronews και θα το κάνουμε και στη συνέχεια, αλλά εγώ θέλω να τονίσω το εξή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση για την ευρωπαϊκή πολιτική. Και αν υπάρχουν λάθη στο τι κάνει το Euronews, ναι, αλλά χτες ακούσαμε ότι πολλά χρήματα χρησιμοποιούνται για τη μετάφραση στο Euronews σε άλλες γλώσσες και αυτό δεν είναι κακό για μένα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε και άλλες γνώσεις που να μην είναι απαραίτητα ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ. Ε, ε, Έχει ζητήσει ακόμα το λόγο ένα συνάδελφος. Θέλει κάποιος άλλος να συμπληρώσει τη λίστα. Όχι, κύριος Βέζερ. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα διαδικαστικό ερώτημα καταρχάς, με κάθε σεβασμό που τρέφω προς το πρόσωπό σας. Ως εκθάματος, Έφτασα στην αρχή της ψηφοφορίας σήμερα το πρωί. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζετε ότι σήμερα το πρωί η κυκλοφορία ε, γύρω από το κυριοβουλίο είναι πραγματικά ε, πολύ ε, έντονη και βαριά και είναι δύσκολο πρόβλημα και δεν είμαι και ο μόνος ευρωβουλευτής που αφήνει το παιδί του στο σχολείο στις 8.30 και παίρνει λεωφορείο για να έρθει στις 9.00. Ε, τα κατάφερα παρόλα αυτά. Σα παρακαλώ όμω να μην οργανώνετε ψηφοφορίες 9 η ώρα ακριβώ, ίσω λίγο αργότερα και να το λάβετε υπόψη σα και εσεί και στη γραμματεία, γιατί δεν είμαι ο μόνος που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα. Είμαι υπέρ. Νομίζω ότι καταγράφονται σωστά οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και η προτεραιότητα ε, και η βούληση της πλειοψηφίας της Επιτροπής μας. Ωστόσο, Θέλω να τονίσω το εξή. Η Επιτροπή δεν λειτουργεί σωστά σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα, κατά τη γνώμη μου. Έχω αποκλίνουσα άποψη σε σχέση με την επικρατούσα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται. Θα έπρεπε να γίνει δομημένο διάλογο με την Επιτροπή, να εμφανιστεί η Επιτροπή, να έχουμε ένα εργαστήριο με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το θέμα, τα πιλωτικά project. Έχουμε πολλά, έχουμε και αντικειμενικά κριτήρια και λέμε ότι υπερψηφίζουμε ορισμένα μόνα, ε, μόνο αυτά τα οποία βαθμολογεί η Επιτροπή με α ή με β έστω. Αλλά είναι υπό και υπό Σε ποια βάζει α και με ποιο τρόπο και γιατί βάζει α σε συγκεκριμένα και σε άλλα όχι. Όλα αυτά δηλαδή είναι μαχητά και υπό συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είναι σωστά προσανατολισμένη η Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν έχει βρει τα κατάλληλα εργαλεία. Νομίζω ότι δεν δίνει την απαραίτητη πολιτική έμφαση που ε, χρειάζεται ε, η στήριξη όλων αυτών των δράσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, σε αυτή την Επιτροπή, χτες δεν είχαμε βέβαια συνεδρίαση, ψηφίζουμε πάντα το πρωί της δεύτερης ημέρας. Ξεκινήσαμε νωρίς, αλλά όχι ακριβώς 9, 9 και 10 ξεκίνησε η ψηφοφορία. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να έρθουν όλοι. Σε αυτή την περίπτωση ίσως ε, μπορείτε να στείλετε τον αναπληρωτή σας εάν είστε σίγουρος ότι θα καθυστερήσετε για τον ένα ή τον άλλο. Πολύ λυπάμαι, καταλαβαίνω ότι έχουμε ο καθένας από εμά δυσκολίες στην προσωπική μας ζωή αλλά ξεκινάει η συνεδρίαση στις 9. Έχω τις ανακοινώσεις της Προέδρου και κατόπιν μετά από 10 λεπτά, γιατί δεν ξεκινάμε ποτέ τις 9 και 10, πριν τις 9 και 10 την ψηφοφορία, αυτό το ξέρετε. Λυπούμε όμως ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις δυσκολίες του καθενός και θα αρχίζουμε την ψηφοφορία 9 και 10. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια για να σας ευχαριστήσω για την στήριξη αυτής της Επιτροπής όσον αφορά τα προγράμματα για την παιδεία και την εκπαίδευση στην αρχή αυτής της νέας θητείας. Σας ευχαριστώ για την πρότασή σας ε, κατά των περικοπών που πρότεινε το Συμβούλιο που θα είχαν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα διάφορα προγράμματα. Κάποια εκατομμύρια στον τομέα του πολιτισμού ξέρετε ότι μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την πρόταση να αυξήσουμε κατά 10% τον προϋπολογισμό του Erasmus ΣΥΝ, ε, το, του οποίου η χρηματοδότηση είχε προβλεφθεί για την τελευταία περίοδο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε πιο επιτυχές πρόγραμμα, μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη κινητικότητα, περισσότερες ε, πρωτοβουλίες, μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ε, και να έχουμε και εγκάρσιους στόχους, ε, δηλαδή να είναι πιο βιώσιμο το πρόγραμμα και να είναι ένα πρόγραμμα για όλους τους πολίτες. Επίσης, θέλω να σε ευχαριστήσω για την στήριξή σας ε, όσον αφορά την πρόταση για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού έρασμους ΣΥΝΑ. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συνέργειες και σε άλλα προγράμματα πολιτιστικά πέρα από το Δημιουργική Ευρώπη και εδώ σκέφτομαι το Ορίζον Ευρώπη ε, ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτά τα προγράμματα και τα διαρθρωτικά ταμεία επίσης. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω πάλι το λόγο στην εισηγήτρια για να μας συνοψίσει αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα σχόλια. Σίγουρα θα φτάσουμε σε ευρεία πλειοψηφία και συνένεση στο τέλος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα συναντηθούμε με τους κοιόδης εισηγητές, θα εμβαθύνουμε κάποια από τα σημεία που χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία και σίγουρα αύριο θα έχουμε τη συζήτηση για το Euronews θα μας δοθούν ε, πιο πλήρεις πληροφορίες, θα ακούσουμε και τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερες ευρωπαϊκές ειδήσει για όλους. Αλλά θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πώς θα το πετύχουμε αυτό. Στην πράξη χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία και συζήτηση το θέμα αυτό και θα δούμε τελικά τι λύση θα επιλέξουμε και για ποιο πράγμα θα συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα σχόλια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με στηρίζετε όσον αφορά τις γενικές μου ε, ιδέες. Είμαστε κατά και των περικοπών του Συμβουλίου, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε ποια είναι αυτά τα προγράμματα που θέλουμε να στηρίξουμε και να προβλα... προβάλλουμε για την επόμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρα. Θέλετε να πείτε κάτι από την Επιτροπή? Thank you very much, uh, Chair. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της DG Connect που είναι υπεύθυνη και για το Creative Europe. Ευχαριστούμε πολύ όσον αφορά τις προτάσεις σας για αύξηση του προϋπολογισμού. Αύριο που θα γίνει η παρουσίαση της έκθεσης του ελεγκτικού Συνειδρίου, βεβαίως και θα συζητήσουμε εις βάθος το θέμα αυτό. Ήθελα να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους για τα θέματα αυτά. Έχουμε εξετάσει εις βάθος το θέμα αυτό και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ουσιαστικά δείχνει ότι μπόρεσε το Euronews με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες και να αναπτύξει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο. Έχουμε ήδη, αν θέλετε, πάρει κάποια μέτρα και κάνει τα πρώτα βήματα για να προχωρήσουμε στην δεύτερη φάση της ανάπτυξης με την σύνθεση όλων των ελέγχων που έχουν γίνει και που γίνονται στην, ε, στο Euronews οι οποίοι θα πρέπει να απλοποιηθούν και να ενοποιηθούν σε έναν μοναδικό έλεγχο. Η επιθεώρηση που έγινε δεν ήταν επιθεώρηση του Euronews αυτού καθεαυτού, αλλά της διαδικασίας εποπτείας του καναλιού. Μπορεί λοιπόν, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει και να σταματήσει κάποιες από τις ε, επαφές που έχει με το Euronews. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για λήξη της σύμβασης, αλλά θέλουμε να εξετάσουμε όλες τις δράσεις που έχουν μέχρι τώρα αναλυφθεί για να υλοποιηθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και πιστεύω ότι αύριο θα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το θέμα αυτό. Και βεβαίως αύριο θα έχουμε μαζί μας και τον ε, κύριο Βιόλα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνο για τα θέματα αυτά. Στις 10 θα έχουμε εδώ μαζί μας ε, τον Υπουργό. Θα διακόψω λοιπόν για 15 λεπτά. Σας παρακαλώ στις 10 ακριβώς να είστε μέσα στην αίθουσα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 12 η ώρα 9 Σεπτεμβρίου. So, ich darf Sie bitten, jetzt wieder Platz zu nehmen. Ich freue mich, die beiden Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ σήμερα να καλωσορίσω θερμά τους δύο Φιλανδούς Υπουργούς, Λι Άντερσον και Χάνα Κόσονεν. Θα μας μιλήσουν για τις προτεραιότητές τους, για τους πολιτικούς ε, άξονες ε, γύρω από τους οποίους ε, θα δημιουργήσουν τα πολιτικά τους προγράμματα που τα οποία θέλουν να μας παρουσιάσουν. Δεν είναι εύκολη εποχή για την Ευρώπη, νέα επιτροπή, Brexit, οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επόμενη περίοδος χρηματοδότησης, ε, το μεσοπρόθεσμο διάστημα της χρηματοδότησης στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και βεβαίως περιμένουμε την φιλόδοξη φιλανδική προεδρία για τομείς όπως η ψηφιοποίηση, η καινοτομία, η έρευνα, η ανάπτυξη, η κατάρτιση, η εκπαίδευση τομείς ε, στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Θέλουμε πραγματικά να στηριχθούν ε, τα βασικά προγράμματα για την κατάρτιση των νέων, για την επαγγελματική κατάρτιση. Θα σας δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο, περίπου 10 λεπτά έχετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε χρόνο για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Νομίζω ότι ότι ο χρόνος ομιλίας που θα δοθεί στα μέλη της Επιτροπής θα εξαρτηθεί από το πόσοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα δούμε επίσης αν ο καθένας θα κάνει την ερώτησή του και θα απαντάτε αμέσως ή αν θα ομαδοποιήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει, η κυρία Άντερσον ή η κυρία Κόσονεν. Έχετε το λόγο κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Εξ ονόματός μου αλλά και εκ μέρους της κυρίας Κόσονεν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να εμφανιστούμε ενώπιον της Επιτροπής σας για να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ και με μεγάλη αγωνία και ενθουσιασμό περιμένουμε και προσδοκούμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η τρίτη Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά άλλαξαν από το 1997 και το 2006 χρονιές κατά τις οποίες είχαμε την Προεδρία για τελευταία φορά. Αυτό είναι αυτονόητο. Ορισμένα πράγματα όμως δεν αλλάζουν ποτέ, παραμένουν τα ίδια. Και κάτι που δεν αλλάζει ποτέ είναι ο φιλανδικός ρεαλισμός κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου. Κάτι άλλο που δεν αλλάζει ποτέ είναι οι καλές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για άλλη μια φορά έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις ήδη στενές θέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Για άλλη μια φορά έχουμε ε, την ευκαιρία να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ένα μέλλον το οποίο θα πρέπει να είναι βιώσιμο από πλευράς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής. Άλλωστε, σύνθημα της ε, Ευρωπαϊκής της Προεδρίας είναι ακριβώς αυτό, μια βιώσιμη Ευρώπη, ένα βιώσιμο μέλλον. Αϊφόρος Ευρώπη, αϊφόρο μέλλον. Οι προτεραιότητες μας είναι οι αξίες, το κράτος δικαίου, η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συμπερίληψη, η κοινωνική ένταξη όλων, η ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλειών και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και η παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές οι προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως υιοθετήθηκε τον Ιούνιο. Ευθυγραμμίζονται επίσης και με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής της ε, κυρίας Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν, έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, σύμφωνα με αυτές τις προτεραιότητες, θα αναπτύξουμε μια σειρά υποπροτεραιοτήτων ανά κλάδο με εύρος και ορίζοντα τα πέντε έτη από πλευράς εκπαίδευσης θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τον πυλώνα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τη σημασία της εκπαίδευσης για όλου, της διαβίου μάθησης, της ε, συνεχιζόμενης εκμάθησης και εκπαίδευσης. Με την Υπουργό κυρία Κόσονεν θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις προτεραιότητές μας σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την εκπαίδευση, οι γενικές προτεραιότητες και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο η οποία θα διευκρινίσει ε, τις προτεραιότητες μας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την, τις επιστήμες, ε, τον πολιτισμό, τα, την άθληση και την νεολαία. Ξεκινώ λοιπόν λέγοντας ότι σημαντικό στοιχείο της Φιλανδικής Προεδρίας το οποίο θεωρούμε ότι συμμερίζεται στο σύνολό του το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρώτον η ανταγωνιστικότητα και δεύτερον η ένταξη όλων, η κοινωνική αν θέλετε συμπερίληψη. Αυτά όλα συμβαδίζουν κατά την άποψή μας. Δηλαδή στο πεδίο των δεξιοτήτων θα επιμείνουμε πάνω σε τρία βασικά σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη ε, σημασία. και βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μας. Πρώτον, θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαβίου μάθηση. Το να μαθαίνει κανείς καθόλου τη διάρκεια της ζωής του για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στις αλλαγές που υφίσταται η κοινωνία, ε, από τις οποίες διέρχεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη μια στρατηγική για διαβίου μάθηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικέ ανάγκες. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη μας προτεραιότητα, θα έλεγα. Να υπάρξει στρατηγική για τη διαβίου μάθηση, γιατί εκεί υπησέρχονται όλα τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, συνοχής και κοινωνικής συμπερίληψης σε ε, ένα κοινωνικό ιστό που υφίσταται ραχδές και συνεχείς αλλαγές. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση συμπληρώνει την έννοια της διαβίου μάθησης, δηλαδή αθρίζει ο άνθρωπος δεξιότητες, εκανότητες, γίνεται, γίνονται πιο ανοιχτά και πιο ευέλικτα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτή η έννοια λοιπόν της συνεχιζόμενης μάθησης ε, καθώς και η έννοια της διαβίου μάθησης λαμβάνει υπόψη της το ρόλο της αλλαγής στη μαθησιακή διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μια πιο ενεργητική δράση για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Πρέπει να δράσουμε και σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικών συστημάτων μας, τα οποία είναι καλό να είναι ανοιχτά να έχουν υψηλό βαθμό συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει τις ίδιες δυνατότητες να μάθει και να συνεχίσει να μαθαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τώρα σε ατομικό επίπεδο τα πολιτικά μέτρα στόχο έχουν να ενισχύσουν την ιδιοκτησία ε, αυτού του προγράμματος. Να ε, το θέλει κανείς να προσυπογράφει σε αυτό το στόχο, ε, να δοθούν σωστές προτεραιότητες και να χαραχθεί σωστή στρατηγική. Και άλλωστε αυτά έχουν, θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης και στο Συμβόλαιο του Νοεμβρίου. Θα γίνει μια πολύ σημαντική, σημαντική συζήτηση τότε, γιατί θα τεθούν οι προσανατολισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εκπαίδευσης. Άλλη προτεραιότητα είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης από σήμερα μέχρι και το 2025. Επιθυμούμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αναπτύξουμε τη διασυνοριακή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιθυμούμε δηλαδή να ενισχύσουμε την μάθηση από ομολόγους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να άρουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο ε, μετά το 2020 και να ενισχυθεί ε, η ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και ε, κατάρτισης και μάθησης. Να αναθερήσουμε τις μεθόδους εργασίας μας, να τις μεταρρυθμίσουμε και να δημιουργήσουμε νέα καινοτόμα εργαλεία και να πρημοδοτήσουμε τα σενάρια που θα βασίζονται στην έρευνα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Άλλη σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης είναι οι θεσμοί, οι φορείς, τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Θέλουμε δηλαδή να, ενθαρρύνουν, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συζητήσουν για αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Και έχουμε αναπτύξει συμπεράσματα που θα πρέπει να ευθετηθούν από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Τώρα για το Erasmus Plus, να σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και θα διαμορφώσει αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης. Το έχουμε διατηρήσει. Έχουμε διατηρήσει και το όνομα του προγράμματος αυτού και αυτό είναι καλό, γιατί ε, ε, περιλαμβάνει πολλές ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ε, του μαθητή, του σπουδαστή. Ξέρετε, το όνομα Erasmus Plus δείχνει ότι είναι ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα το οποίο δεν απευθύνεται μόνο σε όσους βρίσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι οι απόψεις μας συγκλίνουν και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε οικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση αυτή. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, προσυπογράφουν, στηρίζουν ολόθερμα το πρόγραμμα Erasmus Plus. Οι πιο πρόσφατες μελέτες αλλά και διαχρονικά το καταδεικνύουν αυτό ότι είναι το τρίτο πιο σημαντικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα μήνυμα ισχυρό που μας στέλνουν οι πολίτες και πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη να το πάρουμε. Θέλουμε λοιπόν τριμερή διάλογο, τρίλογο για αυτό το πολύ σημαντικό κανονισμό και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Επομένως με ενθουσιασμό μπαίνουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, εάν επιτρέπει η Πρόεδρος, θα ήθελα να έλθω στην τρίτη προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας για τα θέματα αυτά. Για την εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση της έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε το πρώτο συμβούλιο στο οποίο θα συνεδριάζουν Υπουργοί Οικονομικών και Υπουργοί Παιδείας μαζί για να τονίσουμε τη σημασία που έχει η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συμπερίληψη, η κοινωνική ένταξη για όλους. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, αυτό είναι απαραίτητο για την αηφόρο ανάπτυξη, για την ανταγωνιστικότητα, για την προσαρμογή στις κοινωνικές αλλαγές. Όλα αυτά γίνονται μέσα από μια επιωτική εκπαίδευση και μάλιστα για όλους τους πολίτες. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση όντως επιζητούν και απαιτούν την προσωπική ανάπτυξη και αυτό είναι πολύ καλό για να μπορέσει κανείς να καταπολεμήσει τη φτώχεια και να αποφύγει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είμαι στη διάθεσή σας ε, για τα σχόλιά σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Άντερσον, την κυρία Υπουργό. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κώστανον και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι ερωτήσει των μελών. Κύρια Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, όπως και η Υπουργό κυρία Άντερσον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε σήμερα τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Προσβλέπω στην επικοδομητική μας συνεργασία σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα που έφυξε η συνάδελφος, υπουργός, δηλαδή να ξεκινήσω από τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο. Το θέμα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα της Προεδρίας μας για να εξασφαλίσουμε την ισότητα αλλά και την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στην εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στόχος. Η πρωτοβουλία για την νότερη και ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να έχει μια πολύ προσεκτική προετοιμασία χάρη στις ε, εμπειρίες που αποκομίσαμε από 17 πιλωτικά δίκτυα, τα οποία επιλέγησαν τον Ιούνιο, μπορούμε σήμερα να έχουμε ένα προσχέδιο αυτής της πρωτοβουλίας. Πολύ σημαντική είναι λοιπόν και η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία και στις 7 Νοεμβρίου θα γίνει ε, εδώ μια συνάντηση στις Βρυξέλλες όπου έχουμε ε, προσκαλέσει αυτά τα πιλωτικά δίκτυα, τους εκπροσώπους τους, τα κράτη-μέλη και βεβαίως μπορείτε να συμμετάσχετε όλοι. Οι υπεύθυνοι υπουργοί ε, για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση των κρατών μελών θα συζητήσουν ε, επί τη ευκαιρία λοιπόν θέματα που έχουν σχέση με τα πανεπιστήμια και επίσης θα ε, συζητήσουν και όσον αφορά ε, τα πορίσματα που θα υιοθετήσει το Συμβούλιο ε, την επόμενη μέρα όσον αφορά την εκπαίδευση. Τώρα όσον αφορά τον πολιτισμό, είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε ιδιαίτερα το θέμα των ικανοτήτων όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού και τον οπτικοακουστικό τομέα. Και οι προτεραιότητές μας είναι οι εξής. Έχουμε το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027. Αυτή θα είναι και η δική μας προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας. Και είμαι σίγουρη ότι συμφωνούμε όλοι στο ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι η προστιθέμενη αξία και ένα τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης. Ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι λοιπόν απαραίτητος για μια μελλοντική Ευρώπη πιο ισχυρή οικονομικά και χωρίς αποκλεισμούς. και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τον τομέα αυτό και ε, να ε, εξασφαλίσουμε επίσης μια πρόσκοπτη μετάβαση. Όσον αφορά λοιπόν το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε λοιπόν να λάβει πρωτοβουλίες για τη μελλοντική χρηματοδότηση. Η εντολή του Υπουργείου επιβεβαιώθηκε τον Απρίλιο ήταν διαδικασίες οι οποίες διήρκησαν για πολλού, πολλούς μήνες. Ευχαριστούμε λοιπόν την Προεδρία της Αυστρίας και την Προεδρία της Ρουμανίας, τους προκατόχους μας για το επικοδομητικό τους έργο. Και εμείς βεβαίως θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με εσά πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Δεύτερον, εμείς ως Προεδρία θέλουμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ευρώπης για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό μέσω ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου. Ενθαρρύνουμε λοιπόν, παροτρύνουμε την Κομισιόν να καταρτήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική ολοκληρωμένη για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030 μετά από το αίτημα ε, τόσο του Συμβουλίου όσο και του Ευρωκοινοβουλίου. Τρίτον, έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε διαβούλευση για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον οπτικοακουστικό τομέα και να του εμφυσίσουμε νέα πνοή. Θα λάβουμε υπόψη μας τις νέες τεχνολογίες βεβαίως, την καινοτομία σε όλους τους τομείς και την θέση μας στις διεθνείς αγορές. Αλλά ε, θα μεριμνήσουμε και για το περιεχόμενο, τη σχέση μας με το κοινό όσον αφορά την ε, πολυμορφία αλλά και την ισότητα. Όλα αυτά θα τα συμπεριλάβουμε. Επίσης θα προωθήσουμε ένα σχέδιο εργασίας για τον πολιτισμό, το οποίο υιοθετήθηκε ήδη το Νοέμβριο του 2018 και που επιμένει, ε, εστιάζει στις προτεραιότητες του πολιτιστικού και οπτικοκουστικού τομέα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το προσαρμόσουμε στην ψηφιακή, ε, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ε, στα ε, σε από την παγκοσμιοποίηση. Όσον αφορά τώρα την νεολαία, η στόχη μας είναι η εξή. Ποιότητα της εργασίας των νέων, ίσες ευκαιρίες για τους νέους, κατάρτιση για τους νέους εργαζόμενους και τέλος, ψηφιακή εργασία. Ποιοι είναι οι στόχοι μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η κατάσταση νομίζουμε είναι σαφής. Οι θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επ' αυτού, του Ευρωκοινοβουλίου, είναι αρκετά ε, κοντά και θα ξεκινήσουμε λοιπόν διαβουλεύσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. οι νέοι εργαζόμενοι, είτε επιπληρωμή είτε εθελοντικά, θα πρέπει να έχουν τις ανάλογες ικανότητες και να μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να βρούμε μέτρα και να εφαρμόσουμε ε, μία μέθοδο βιομοτήμων. Και βεβαίως εδώ θα ε, ε, ε, ζητήσουμε από το Συμβούλιο να εκδώσει συμπεράσματα επ' αυτού. Τώρα όσον αφορά την ψηφιακή εργασία των νέων. Υπάρχουν δυνατότητες και αυτές οι δυνατότητες και ευκαιρίες θα πρέπει να είναι οι ίδιες για όλους. Να ενισχύσουμε, θέλουμε, εδώ τις ψηφιακές ικανότητες και οι νέοι να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνίες που γίνονται όλο και πιο ψηφιακέ και τεχνολογικές και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα και σε αυτό θα ζητήσουμε επίση από το Συμβούλιο να εκδώσει συμπεράσματα. Όσον αφορά τον τομέα του αθλητισμού, δύο είναι οι προτεραιότητές μας. Καταρχάς, η πάλι κατά της διαφθοράς. Είναι μία από τι προτεραιότητε τη προεδρία μα. Θέλουμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική αποτελεσματική όσον αφορά την πάλη κατά της διαφθοράς. Και αυτό θα το κάνουμε μέσω ενός προβληματισμού, μακροπρόθεσμου, αλλά και μέσω της άριστης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφανή διακυβέρνηση και αυτό σε όλους τους τομείς του αθλητισμού. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά την σύμβαση Μακόλιν προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επικύρωσης εκ μέρους των κρατών μελών και θα πρέπει να εργαστούμε ένεργα επίσης και για την πάταξη του ντόπινγκ. Άλλη προτεραιότητα, η, η προστασία των παιδιών και των νέων στον τομέα του αθλητισμού. για κάθε άθλημα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται ε, με το συγκεκριμένο άθλημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά και τους νέους. Τέλος, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας πρόσκληση. Ελπίζω ότι οι διοργανικές μας σχέσεις ε, θα αποδώσουν καρπούς και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Μας έθεσαν με σαφήνεια το επίκεντρο και τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στους συντονιστές για δύο λεπτά στον καθένα. Και κατόπιν θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μέλη. Θα δούμε ανάλογα με το πόσοι θα εγγραφούν στη λίστα των ομιλητών σας παρακαλώ δείξτε ποιος θέλει να πάρει το λόγο για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Ξεκανώ με την Μιχαέλα Σόντροβα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις δύο υπουργούς ε, για τις παρουσιάσεις τους. Εδώ βρίσκεστε ενώπιον μιας επιτροπής που ασχολείται με τον πολιτισμό και έχουμε πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες από την Φιλανδική Προεδρία. Όλοι ξέρουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήθελα να σας κάνω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις για το Εράσμους. Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε να το στηρίξετε, να το διατηρήσετε και να το στηρίξετε και ελπίζω ότι αυτό θα ακολουθηθεί και από μια αύξηση του προϋπολογισμού για το 2020 αλλά και περαιτέρω στηρίξη στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή μας μίλησε για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του Εράσμους. Μια δηλαδή σημαντική αύξηση. Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν όλα αυτά τα ποσά. Εσείς μιλήσατε για την κάλυψη των αναγκών όλων των σπουδαστών. Για μας αυτό είναι ο στόχος μας. Σήμερα φυσικά αυτό δεν συμβαίνει. Δεύτερον, όσον αφορά την προετοιμασία του επόμενου οικονομικού έτους, κοινός μας στόχος είναι να πατάξουμε την παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσει, το λαϊκισμό, τη δημαγωγία και το Εράσμους θα μπορούσε να επιληφθεί και αυτών των τομέων. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που έχουμε δύο υπουργούς εδώ μαζί μας, έναν αρμόδιο για την παιδεία και έναν για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για όλες σας τις προσπάθειες για να πείσετε τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τη χρηματοδότηση. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Είναι σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον εθελοντισμό και που θέλουμε να στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άντερσον, ευχαριστώ πολύ κυρία Σόεντροβα για την ερώτησή σας. Εγώ θα απαντήσω για το Εράσμους και η συνάδελφος θα μιλήσει για το Σώμα Αλληλεγγύης. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, το Erasmus Plus είναι ένα πολύ γνωστό, ίσως από τα πιο γνωστά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι για μας ε, μια καθοριστική προτεραιότητα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο και τις διαπραγματεύσεις για αυτό το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ακόμα εκρεμή θέματα, όπως αυτά που αφορούν τα δημοσιονομικά και τα οποία είναι εκτός των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι θέμα και αρμοδιότητα της τελευταίας φάσης, δηλαδή το αναλαμβάνουν οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων μετά το πέρας των υπόλοιπων διαπραγματεύσεων. Βεβαίως ε, οι τεχνικές πτυχές θα ρυθμιστούν κατά την άποψή μας, ήδη έχουν βρεθεί στις τεχνικές συναντήσεις πολύ ικανοποιητικές συμβεβαστικές λύσεις. Κάποια ακόμα θέματα ε, χρήζουν περαιτέρω συζήτηση και αυτό θα γίνει στον τριμερή διάλογο. Όπως παραδείγματος χάρη και αυτό θα είναι αντικείμενο του τριμερούς διαλόγου, είναι η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, η ενσωμάτωση όλων, η, η κινητικότητα ατόμων ε, ενηλίκων και βεβαίως ό,τι έχει σχέση με τον ε, αθλητισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα είναι προτεραιότητες και θα στηριχθούν από την Προεδρία της Φιλανδίας. Η κυρία Κόσοβα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστώ. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και οι παρατηρήσεις. Ε, και εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να στηρίξουμε την πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν κοινά σημεία με το Εράσμος και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε και να δείξουμε στους νέους Ευρώπης ότι υπάρχουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Η Πέτρα Κάμερβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ θερμά τις δύο υπουργούς. Πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, αντιλαμβάνομαι από τις παρουσιάσεις σας, γιατί ουσιαστικά σας μένουν ακόμα τέσσερις μόνο μήνες. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και θα διασφαλίσουμε την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά μας. Όσον αφορά το Erasmus και το Erasmus Plus, είναι όντως στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών ένα από τα πιο εμφανή και φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράμματα. Για το 20 αποφασίσαμε ότι και όσον αφορά το Εράσμους αλλά και όλα τα άλλα προγράμματα δεν θα δεχθούμε τις ε, περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο. Εμείς μάλιστα προτείνουμε συν 10% για το Εράσμους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη της Φιλανδικής Προεδρίας και βεβαίως σας εύχομαι κουράγιο γιατί πρέπει να πείσετε όλους τους υπόλοιπους υπουργούς, τους αρμόδιους για τα θέματα χρηματοδότηση αυτών των ε, προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές οι πρωτοβουλίες που αναλάβατε μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει τα λόγια να ακολουθηθούν από πράξη. Επαναλαμβάνω γιατί ξέρω την κατάσταση ότι δεν είναι εύκολο να πείσουμε τους Υπουργούς Οικονομικών για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Μιλήσατε για την ε, διαβίου και τη βιώσιμη, την ε, διαβίου κατάρτιση και την ε, συνεχή κατάρτιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι εδώ συμφωνεί και η Επιτροπή, θα στηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Δυστυχώς αμφιβάλλω αν αυτό θα το κάνουν πολλά κράτη-μέλη. Όπως είπε η συνάδελφος Σόιντροβα, η Φιλανδία αποτελεί τρανό παράδειγμα στους τομείς αυτούς. Και βεβαίως σήμερα βλέπουμε ότι όλο και πιο πολύ στοχεύουμε στις δεξιότητες, τα skills. Ίσως θα πρέπει να θέσουμε κάποιους κοινού στόχους προηγουμένως και κατόπιν να δούμε ποιος είναι σε θέση να τους υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο ή από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ας είμαστε ρεαλιστές, ας θέσουμε κοινούς στόχους που να μπορεί να υλοποιηθούν και κατόπιν θα δούμε ποιος. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία. Θέλετε να απαντήσετε, κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάμερβερτ, για τις ερωτήσεις σας. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο. Η Φιλανδοί όμω είναι γνωστή για την αποτελεσματικότητά του και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα για την ε, από κοινού συνεδρίαση Διευρυμένου Υπουργικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Υπουργών Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή Υπουργών Οικονομικών και Υπουργών Παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε μαζί για να τονίσουμε τη σημασία τη επένδυση στην εκπαίδευση, επένδυση στην έρευνα. Επένδυση στην εκπαίδευση και στην έρευνα για λόγους ισότητας, αλλά και για λόγους οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει αυτό να το τονίσουμε και να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Τώρα, ως προς το Erasmus Plus, επαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ στοχοπροσυλλομένοι. Μας ενδιαφέρει να ξεκινήσει ο, τριμερό, ο τριμερής διάλογος, οι διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα. Ο προπολογισμό είναι πρόβλημα που πρέπει να ρυθμιστεί αργότερα γιατί επηρεάζεται ιδιαίτερω από τι διαπραγματεύσει για το συνολικό ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, για εμάς είναι σημαντικό να εργαστούμε μαζί με εσάς, να συνεργαστούμε με εσάς, να συνεργαστούν τα δύο θεσμικά όργανα και τα τρία ε, ε, για τα θέματα που μας απασχολούν και τους τρεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ministerin haben Sie noch? Η Υπουργό Κόσονεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας για τις εξαιρετικές αυτές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Κάμερβερτ για την τοποθέτησή της. Κοιτάξτε, ως προς την επικουρικότητα πρέπει να θέσουμε κοινό στόχο και ίσως αυτή είναι και η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα για την επικουρικότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεγόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ τις αξιότιμες ε, κυρίες ε, υπουργού για την ε, παρουσίαση τους και την παρουσία τους εδώ. Προσυπογράφω πλήρως αυτά τα οποία είπατε για την ψηφιακή εκπαίδευση, για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για την ε, βιομηχανία της δημιουργίας, του θεάματος και του πολιτισμού, αλλά και ό,τι είπατε για τη συνεχιζόμενη και διαβίου μάθηση. Η λέξη πολιτισμός δεν αναφέρονταν στο κείμενό σας, αλλά προφορικά μας διαβεβαιώσατε και μας καθησυχάσατε και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερως. Ε, με ενδιαφέρει όμως και η μαθησιακή διαδικασία και η μάθηση ε, στον τομέα των, της βιοτεχνίας, ε, των, ε, της εξειδίκευσης ως μέσο καταπολέμησης της ανεργίας μεταξύ άλλων. Εμείς θέλουμε να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός στο Erasmus Plus και πρέπει να συμπεριλάβει και αυτού του είδους την εκπαίδευση. Να υπάρχει μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γίνεται ήδη αυτή η δουλειά και είναι σημαντική. Θέλω να τονίσω και το θέμα του πολιτισμού και της ε, κουλτούρας, δηλαδή την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, είτε σε υλικό επίπεδο, την ανάδειξη δηλαδή των κτηρίων και μνημείων που συγκροτούν την ιστορία μας, αλλά και την άλλη άειλη κληρονομιά μας και κυρίως την γλωσσική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φαράγκ για τις ερωτήσεις σας. Χαίρομαι που ε, ακριβώς αναφερθήκατε στην ε, περιστασιακή κατάρτιση και εκπαίδευση, την επαγγελματική, συγγνώμη. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την κατάρτιση και στο πλαίσιο του έρασμους ΣΥΝ, τώρα και στο μέλλον. Η Φιλανδία Θέλει λοιπόν να προωθήσει την επαγγελματική κατάρτιση. Θέλουμε να είναι μια πολύ καλή ελκυστική επιλογή για τους νέους φοιτητέ, για να έχουν ποιοτικέ εργασίες στο μέλλον και για να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους. Επίσης, θέλουμε να είναι ίση ε, με την ανώτερη και, ε, ανώτερη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να μην υπάρχουν δηλαδή ε, εδώ διαφορές και να, μπορεί έτσι, ε, να, ε, να μπορούν έτσι όλοι αυτοί οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλες σπουδέ. Να έχουν επιλογές, να μπορούν δηλαδή να συνεχίσουν τις σπουδέ τους και σε ακόμα ανώτερο επίπεδο στη συνέχεια. Νομίζουμε λοιπόν ότι μια ποιοτική επαγγελματική ε, κατάρτιση μπορεί να ε, μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη προβολή ως Ευρώπη, ότι είναι μια Ευρώπη η οποία ε, παρέχει δεξιότητες και θα ε, κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο Ελσίνκι για την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Προεδρίας μας και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία ούτως ώστε να δημιουργήσουμε προβολή. Μια θετική προβολή λοιπόν για την επαγγελματική κατάρτιση. η Κορσόνεν. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Το 2018 ήταν το έτος πολιτισμού και όπως ξέρετε για μας ο πολιτισμός είναι προτεραιότητα. Και όπως είπατε, και επανέλαβαν και οι αρχηγοί κρατών. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την ιδέα του ε, έτους πολιτισμού. Και στο πρόγραμμα εργασιών της Προεδρίας αναφέρεται ο πολιτισμός. Το 2019 είναι η πρώτη χρονιά όπου εφαρμόζουμε ακριβώς αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον πολιτισμό. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εργασιών με πέντε θεματικές προτεραιότητες. Μιλάμε για την αηφορία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για παράδειγμα. Και είναι ακριβώς αυτή η αηφορία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και ε, από κοινωνικής αλλά και οικονομικής απόψεως, διότι ο πολιτισμός είναι ε, η μεγαλύτερη πηγή πλούτου μας εδώ στην Ευρώπη. Και ως Προεδρία θα επιμείνουμε λοιπόν σε αυτό και θα εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα εργασιών. Σας ευχαριστώ. Στον κατάλογο έχω την κυρία Άντερσον σαν ε, τον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κύριε Υπουργή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, αλλά και για την παρουσίαση των πολύ φιλόδοξων προγραμμάτων Βεβαίως ε, η διασύνδεση των νέων με όλα αυτά τα προγράμματα είναι κάτι που όλοι το επιθυμούμε και το στηρίζουμε. Έχω μία ερώτηση που αφορά την έννοια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αναρωτιέμαι λοιπόν και αυτό αφορά η ερώτησή μου. Έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι κατά κάποιο τρόπο εις βάρος της πολυμορφίας των ε, πολιτισμών μας, ε, των λαών μας και δεν ξέρω αν ε, θα στήριζα μία προσπάθεια ή κάτι που κατά κάποιο τρόπο περιορίζει, συρρυκνώνει αυτήν την τεράστια πολυμορφία των πολιτισμών των ευρωπαϊκών λαών. Δεν ξέρω δηλαδή ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, αυτής ενδυνάμωσης της έννοιας του ευρωπαϊκού πολιτισμού επί της πολυμορφίας και του πολιτισμικού πλούτου που σήμερα γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Πώς το βλέπετε αυτό. Kysymys on tietenkin. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Näitä huolia σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Εννοείται ότι κάθε χώρα μας έχει τον πολιτισμό της, την ταυτότητά της και την πολιτιστική της κληρονομιά. Εγώ δεν βλέπω απολύτως καμία αντίφαση μεταξύ του προγράμματός μας και της στήριξη της πολυμορφίας. Βεβαίως και πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε ο καθένας τον δικό του πολιτισμό. Υπάρχει όμως και ένας κοινό ευρωπαϊκός πολιτισμός, υπάρχουν κοινέ ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες στηρίζουμε. Θα ήθελα να υποθυμίσω ότι η έννοια, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ε, πολιτιστικής, αν θέλετε, προσπάθειας είναι να είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας. Δηλαδή είμαστε Ευρωπαίοι χωρίς αυτό να υπονομεύει και να σβήνει τις δικές μας πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Σας ευχαριστώ. λέει ο κύριος Φραντς. Βεβαίως και είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ευρωπαϊκή πολυμορφία. Σήμερα μιλάμε για το Erasmus Plus, το οποίο επιτρέπει και δίνει την ευκαιρία σε άτομα τα οποία πολλές φορές είναι αντικείμενα διακρίσεων, όπως παραδείγματο χάρη ρατσισμού κατά των τσιγκάνων. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα διακρίσεις και κατηγορίες νέων που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα όπως το Erasmus Τι θέλετε να κάνετε έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus ακόμα και σε αυτούς τους νέους που σήμερα ανήκουν στις κατηγορίες που αποκλείονται. Ευχαριστώ κύριε Φραντς, για τις ερωτήσεις σας. Ως προς την ένταξη ε, και το πρόγραμμα Erasmus Plus, πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό είναι να ε, αναπτύξουμε δομές έτσι ώστε όλοι να συμμετάσχουν στο Erasmus Plus, για όλους να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να είναι ανοιχτό, να είναι διαθέσιμο, να μπορούν οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες, νέοι φοιτητές, οι μαθητές να το κάνουν, ανεξαρτήτως ε, κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου των ιδίων ή της οικογένειάς τους. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για εμάς. Και όπως ανέφερα και νωρίτερα, για το πρόγραμμα Erasmus Plus, πιστεύουμε ότι η ένταξη ε, η κοινωνική συμπερίληψη, το να μην είναι κάποιος απ' έξω, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του τριμερούς διαλόγου, του προβληματισμού μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλος του προγραμματός μας και θέλουμε να το αναπτύξουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ευχαριστώ. Äh, ist äh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ τις δύο υπουργούς. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γνωρίζω την φιλανδική αποτελεσματικότητα. Σας εμπιστεύομαι πλήρως και σας εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο έργο σας. Πώς αντιμετωπίζουμε όμως ορισμένα ζητήματα όπως το εξής. Όταν υπάρχουν σε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαινόμενα ρατσισμού, εθνικισμού, μυσαλλοδοξίας, και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες αρκε... ευρωπαϊκές χώρες ή και αρκετές. Και τελικά έτσι παράγεται λόγος ξενόφοβος ε, που προκαλεί διακρίσεις. Αυτό είναι θέμα. Υπάρχει σε κάποιες χώρες περισσότερο, σε άλλες λιγότερο. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι η εθνική εκπαίδευση συχνά στρέφεται εναντίον ε, της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη ή δεν συμπεριλαμβάνει όλους, εν πάση περιπτώσει, τρόπον τεινά. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό προς συζήτηση. Δεν ξέρω, έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Σας απασχολεί. Ministerin Anderson η Υπουργός κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ κύριε Κίζελ για το ερώτημα αυτό. Είναι ακαθόδες το ζήτημα γιατί είναι και θέμα αρμοδιοτήτων. Αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ε, μιλούμε για το περιεχόμενο βεβαίως της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει, να συντονίσει και να εφαρμόσει δράσεις των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και με αυτή την περιορισμένη αρμοδιότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά μπορεί να κάνει πολλά για να διευκολύνει την ανταλλαγή των ιδεών, τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι Όλα αυτά συνοψίζονται στο ευρύτερο ερώτημα του πώς βλέπουμε το ρόλο της εκπαίδευσης γενικά. Ποιο ρόλο έχουν τα εκπαιδευτικά ε, συστήματα στη διαμόρφωση των κοινωνιών. Δηλαδή, ε, προσωπικά πιστεύω ότι ε, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι το εξής, ότι είναι σημαντικό να έχουν όλοι δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση. Όλο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, αλλά και για την ισότητα και την ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη και άνθηση, αν θέλετε, όλων των πολιτών στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για την πολιτική, για το ρόλο που έχει εκπαίδευση στην πορεία μιας κοινωνίας και στις αξίες που τη διαμορφώνουν. Ευχαριστώ. κυρία Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για αυτό πολύ επίκαιρο ερώτημα. Οι αρμοδιότητες της κάθε χώρας ε, για την εκπαίδευση είναι μεγάλες και η δική σας επιτροπή εδώ μπορεί να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές και να ε, γνωστοποιήσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και οι αρμοδιότητές σας διαπιστώνουμε ότι είναι η καλύτερη κατανόηση των μεν από τους δε. Όντως υπάρχει μια μεγάλη πολυμορφία πολιτιστική και πρέπει οι διαφορές να γίνονται γνωστές. Νομίζω ότι ένα τρανό παράδειγμα αυτού είναι και το Erasmus Plus. Για μας λοιπόν, μέσω του Erasmus Plus συνειδητοποιούν οι νέοι πώς ζουν και πώς μπορούν να ενδυναμωθούν γνωρίζοντας νέες πραγματικότητες. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους νέους και έχουμε αρκετά συστήματα που προωθούν αυτές τις ιδέες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τον γύρο των εισηγητών και μπορούμε να περάσουμε στα μέλη της Επιτροπής. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχουμε πάρα πολλά ονόματα στον κατάλογο, να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, η Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά τον τριμερή διάλογο για το Erasmus ΣΥΝ. Θα μπορούσαμε λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου. Ε, θα ήταν κάτι που θα θέλαμε. Ε, ε, λοιπόν, θα συγκεντρώσουμε δύο ερωτήσεις για να απαντηθούν από κοινού. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριος Ρουίθ Τεμπέσα. Θέλω να ευχαριστήσω τις δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις τους, πολύ ε, συγκεκριμένες. Καλό θα ήταν να μην ήταν, να ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένες, γιατί ήταν κάπως γενικόλογες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα βρούμε, δεν πειράζει. Δεν αναφερθήκατε όμως καθόλου και φαίνεται να μην είναι δικιά σας προτεραιότητα η εκπαίδευση στην έννοια της ε, και στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας αν θέλετε. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα πρέπει να το συμπεριλάβατε αν σας έχει περάσει καθόλου από το μυαλό αυτή η σκέψη ή δεν μπορέσατε να το συμπεριλάβατε ενώ το έχετε σκεφτεί. Η συντονίστρια Κέα Κάμερβερτ και άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερως είναι οι περικοπές που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια και για του χρόνου για το πρόγραμμα Creative Europe. Αυτό μας ανησυχεί. Και από ό,τι ξέρουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλει να επιβάλλει περικοπές σε αυτό και θέλει να επιβάλλει περικοπές και στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Ε, οι δύο υπουργοί μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν αυτό, η κυρία ε, Κόσον και η κυρία Άντερσον. Είναι αυτή η θέση του Συμβουλίου και αν ναι, αντιτάσσονται ορισμένα κράτη-μέλη σε αυτή την ε, άποψη που είναι υπέρ των περικοπών και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Όπως γνωρίζετε, η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος ειστερεί κατά πολύ συγκριτικά με το πρόγραμμα Εράσμος. Και αφού προτείνουμε την αύξηση του προπολογισμού για το Εράσμος, δεν μπορούμε να κάνουμε και μια επιπρόσθετη προσπάθεια ε, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ οι δύο υπουργοί μπορούν να απαντήσουν. Ζητώ συγγνώμη, ναι, είχατε ζητήσει το λόγο πιο νωρί, αλλά θα πάρετε το λόγο αμέσω. Δίνω όμω αμέσω το λόγο στου δύο υπουργού για να απαντήσουν στι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω απαντώντας τον κύριο Σβέρ, διαπραγματεύσεις για το Erasmus Plus. Όσον αφορά το πρόγραμμα, είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν το τέλος του χρόνου. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση όμως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Εν ώψη του Brexit και άλλων ενεξελίξη καταστάσεων, Θεωρούμε ότι είναι μάλλον απίθανο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντεμπέζα για τις ερωτήσεις που έκανε όσον αφορά την εκπαίδευση, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες. Ναι, ο ρόλος που παίζει η εκπαίδευση των νέων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες είναι καθοριστικό και βεβαίως το Σώμα Αλληλεγγύης και το Erasmus Plus δίνουν στους νέους της Ευρώπης μια δυνατότητα να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, να ταξιδέψουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωρίσουν νέες συνήθειες. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν και η δουλειά που κάνουμε εμείς στη Φιλανδία είναι πολύ κοντά στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών. Η κυρία Κόσονεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Η δημιουργική Ευρώπη με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Και βεβαίως το Συμβούλιο πρότεινε τη μείωση των ποσών που έχουν προταθεί από την Επιτροπή και αυτό αφορά όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού αλλά και την Δημιουργική Ευρώπη. Βεβαίως πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη στάση των κρατών στο Συμβούλιο. Υπάρχουν οι χρηματοδότες και υπάρχουν οι αποδέκτες των κονδυλίων και της χρηματοδότησης. Βεβαίως, ο τελικός προϋπολογισμός θα συναποφασιστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε στην αρχή της διαπραγμάτευσης που αφορά τα δημοσιονομικά και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της διαδικασίας που ελπίζουμε να φτάσει στην τελική της φάση στο τέλος του χρόνου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η διαπραγμάτευση αφορά όλα τα προγράμματα και θα δούμε τι θα γίνει συγκεκριμένα με τα συνολικά ποσά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, σαν συντονίστρια, θα πάρει το λόγο η κυρία Μεμπάρτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του ECR θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις δύο υπουργούς, την κυρία Κόσονεν και την κυρία Άντερσον, για τις παρουσιάστες. Πολύ ισορροπημένη και φιλόδοξη παρουσίαση και πρόγραμμα Όντως, η Φιλανδία έχει μεγάλες επιτυχίες και όσον αφορά την καινοτομία και όσον αφορά το εκπαιδευτικό της σύστημα. Και βεβαίως σας συγχαίρουμε όλοι και θαυμάζουμε το πρόγραμμα της διαβίου και της συνεχούς κατάρτισης που προτείνεται για τους νέους της χώρας σας. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η πτυχή της ε, στρατηγικής που αφορά την τέχνη Επίσης, μία άλλη ερώτηση που αφορά την ολοκληρωμένη ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το θέμα των μέσων, των οπτικοακουστικών μέσων, των πολυμέσων, όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη ασφάλεια. Δεν άκουσα τίποτα για τον τομέα αυτό, αλλά μιλήσατε για τρία διαφορετικά μέσα είναι ένα θέμα που σίγουρα θα συζητηθεί εκτενέστατα μεταξύ των Υπουργών ε, στο Συμβούλιο. Κυρία Κόσονεν. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Μερικές φορές πρέπει να συζητήσουμε ποιος είναι αρμόδιος, γιατί πριν να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Αναφέρατε πρώτα-πρώτα την συνεχή μάθηση, ε, ένα από τα θέματα που θέλουμε να τονίσουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας και νομίζω ότι αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε για την ολοκληρωμένη ασφάλεια. Για μας ε, η ανάγκη για συνεχή μάθηση απορρέει από τις τεχνολογικές εξελίξεις, από την ψηφιοποίηση, την, την αυτοματοποίηση στο, στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τόσο ο καθένας χωριστά, όσο και όλη η κοινωνία, να έχουμε τα μέσα να ε, προσαρμοστούμε σε αυτές τις εξελίξεις. Και αυτό συνδέεται και με τις ψηφιακές δεξιότητες. Να μπορούμε δηλαδή, να μπορούν τόσο οι νέοι ε, μαθητές, ε, όσο και οι μεγαλύτεροι, να βελτιώσουν και να εξυγχρονίσουν τις δεξιότητές τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε αυτή την ολοκληρωμένη ασφάλεια. Αλλά είναι επίσης σημαντικό ε, όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσει, τα fake news που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική που θα επιλέξουμε για αυτά. Υπουργό Κυριακό Σόνεν. Ευχαριστώ για αυτές τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Όσον αφορά την θέση της Φιλανδίας για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη, η παιδεία όσον αφορά στον τομέα της μουσικής είναι, έχει αξία 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η θέση μας από αυτού. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι στο επίκεντρο ε, των δράσεών μας. Και θα έλεγα ότι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον τύπο. Θα πρέπει να έχουμε ένα θεματολόγιο όμως όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επίσης όσον αφορά την εξοικείωση, την παιδεία, όσον αφορά τα μίντια. Αυτό θα κάνουμε και στον τομέα της παιδείας και έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές ε, που υπάρχουν και να ε, προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους. Ο κύριος Μοχάμετ ο κύριος Φραντς είναι η επόμενη. Δεν είναι εδώ. Εγώ είμαι πρώτος. Πριν αναφέρατε το Brexit και μιλήσατε για μείωση του προϋπολογισμού, υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα διοργανώσετε όσον αφορά το Brexit και όσον αφορά την συνεισφορά σε όλη την Ευρώπη. Εγώ αποσύρω την ερώτησή μου γιατί απαντήθηκε ήδη. Ο κύριος Φραγκόσκι λοιπόν. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za prezentację priorytetów prezydencji. ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Μία ερώτηση για τον αθλητισμό θα ήθελα να κάνω. Η προστασία των παιδιών στις αθλητικές διοργανώσεις. Μπορείτε να μας δώσετε απτά παραδείγματα μέτρων. Τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η Προεδρία της Φιλανδίας στον τομέα αυτό. Ποιος θέλει να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Uh, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μοχάμεντ ε, για το θέμα του Brexit, την ερώτηση σχετικά με το Brexit. Γενικά, η προτεραιότητά μας ως Προεδρία είναι να υπερασπιστούμε την ενότητα, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως Προεδρία είμαστε αφοσιωμένοι στην γραμμή που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι υπέρ της... Έχει μια συμφωνία μάλλον απόσυρσης και όσον αφορά την επιτροπή αυτή, όσον αφορά το έρασμος ΣΥΝΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο σε οποιαδήποτε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία αποχώρηση θα συμμετέχει κανονικά και εάν υπάρξει τελικά συμφωνία αποχώρηση, θα συνεχίσει να συμμετέχει κανονικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Αλλά αν φύγει χωρί συμφωνία, ε, τότε ε, μπορεί να υπάρξουν κάποιες ε, δράσεις κινητικότητας, αλλά βεβαίω όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά το πρόγραμμα θα λήξουν με την αποχώρηση. Η Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας, κύριε Φανκόσκη. Όσον αφορά την ασφάλεια των νέων και των παιδιών στον αθλητισμό, πρέπει να βασιστούμε στην, ε, μάλλον βασιζόμαστε στην εργασία μέχρι τώρα και αυτό που θέλουμε να κάνουμε ε, βασίζεται στα πορίσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την ασφάλεια των νέων και των παιδιών. Στόχος μας είναι, πολύ απλά, να ε, δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιε οι προκλήσεις και να εξετάσουμε κάποιε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βελτίωση της ασφάλειας. Τα, πορά, του Συμβουλίου έλεγαν ότι πρέπει να αυξήσουμε την ασφάλεια ε, στον αθλητισμό για τα παιδιά και τους νέους, όπως επίσης και για την υγεία τους στις 24 Σεπτεμβρίου έχουμε προβλέψει να κάνουμε ένα συνέδριο από ε, αυτού του θέματος. Σμερίλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπούντιν και μετά κύριο Σμερίλιο. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, για την επέκταση του Erasmus για να περιλάβει και όσους κάνουν στάζ, όσους ε, διανύουν περίοδους μαθητείας. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και την προσυπογράφω. Δύο σχόλια. Πρώτον, πρόσκληση. Σας καλώ... Έχω καλέσει στις 16 Οκτωβρίου μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν στάζ έτσι ώστε να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να έχουν ένα, μια εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί με το Brexit και θέλω να σας καλέσω ε, στην ε, συνάντηση που θα έχουμε με αυτούς και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Από εκεί και πέρα θέλω να μιλήσω για τα βραχυχρόνια συμβόλαια ε, νέων ανθρώπων που δουλεύουν στο οπτικοακουστικό τομέα και αλλού με λιγότερες ευκαιρίες νέοι και λιγότερη εκπαίδευση. Τι προτίθεστε να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάσει ο κόσμος την, το όραμά του, δεν θα παχυδευτεί σε αυτή την αέναη προσωρινή απασχόληση ε, για να έχει μια κάποια κοινωνική προστασία και μια κάποια κοινωνική κινητικο, και εργασιακή κινητικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, επίσης για τη συμβολή σας. Νομίζω ότι εμείς χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο. Ε, μια ανάπτυξη που να βασίζεται στην παιδεία, την γνώση και τον, ε, και τον πολιτισμό. Και σκέφτομαι κυρίως την δημιουργική Ευρώπη. Είχαμε μια άριστη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειαζόμαστε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η έχουμε μια, ήδη μια μακρά εμπειρία. Θα πρέπει λοιπόν να την εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπειρία και να βελτιώσουμε το πρόγραμμα, να το κάνουμε πιο απλό, πιο διαφανές και να ε, έχουμε μεγαλύτερη προβολή ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, να εργαστούμε όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων, ε, να έχουμε μια εξακρίβωση εκ των υστέρων του κατά πόσο το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη είναι αποτελεσματικό και επ' αυτού θα ήθελα να τονίσω ότι είναι αλήθεια. Ο πολιτισμός βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του εξαμήνου εργασιών αλλά είναι και το θέμα της χρηματοδότησης, πολύ σημαντική για όλα μας τα προγράμματα, ακόμα πιο σημαντική όμως για την Δημιουργική Ευρώπη. Um, Ευχαριστώ. Να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Μπέντιν πρώτα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα περιμένουμε να τη λάβουμε με ιδιαίτερη ε, χαρά για την εκδήλωσή σας στις 16 Οκτωβρίου. Πώς θα εργαστούμε για την κοινωνική κινητικότητα, για να μην χάσουν τις ελπίδες τους οι νέοι φοιτητές, μαθητές, νέοι άνθρωποι που ενδεχομένως δεν έχουν εκτεταμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και μεγάλη εκπαιδευτική διαδρομή. Το πιο σημαντικό είναι να συμπεριλάβουμε αυτή την έννοια της ένταξης σε όλες τις εκπαιδευτικές ε, πολιτικές. Το καλύτερο όπλο ε, κατά της απομάγευσης αν θέλετε, της απώλειας των ελπίδων είναι η, η, η συμμετοχή, η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα ποιοτικό που λαμβάνει υπόψη του τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν όλες τις χώρες. Να υπάρχουν δυνατότητες, για παράδειγμα, για όλες τις οικογένειες και για όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση από νωρίς στη ζωή τους σε εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας. Τον λέω αυτό διότι γνωρίζω πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες με τη μετανάστευση και η υψηλή ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει. Ε, σε κάθε περίπτωση εμείς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση στην ε, πολύ νεαρή παιδική ηλικία και η φροντίδα σε αυτές τις ηλικίε, ε, ιδιαίτερο των παιδιών που έρχονται από χαμηλότερο κοινωνικό υπόβαθρο, είναι απολύτως απαραίτητη, είναι καθοριστική σημασίας. Και ε, η υψηλή ποιότητα σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους να συνεχίσουν τις ε, σπουδές τους στη συνέχεια εφόσον το επιθυμούν, να μην υπάρχουν κλειστές πόρτες δηλαδή, αλλά να είναι συγκοινωνούντα δοχεία ε, οι διάφορες εκπαιδευτικές διαδρομές, τα εκπαιδευτικά συστήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόσονεν. Σας ευχαριστώ κύριε Σμερίλιο, δεν προφέρω σωστά το όνομά σας και λυπούμε πολύ γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Συμφωνώ πολύ με τα λεγόμενά σας για το στόχο του προγράμματος και θα το στηρίξω με μου τις δυνάμεις, ξέρετε. Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Ένα λεπτό. Μπλάνκο και Πόλακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις δύο υπουργούς για την παρουσίαση του προγράμματος της Φιλανδικής Προεδρίας που όντως είναι φιλόδοξο πρόγραμμα. Εγώ δεν γνωρίζω τη φιλανδική αποτελεσματικότητα, αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας. Λίγο λίγα έχουν υποθεί για τη σημασία του πολιτισμού και για τη θέση που έχει ο πολιτισμό στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων τη Φιλανδική Προεδρία. Εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία αυτού. Δε, όχι για να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπάρχει ευρωπαϊκό πολιτισμό και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσαρκώνει ε, το απάβγασμα των ε, ευρωπαϊκών αξιών, αν θέλετε. Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την τη συνειδητοποίηση όλων ότι μοιραζόμαστε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και βρίσκεται μέσα μας και το μοιραζόμαστε όλοι. Ως εκ τούτου, ε, θέλω να τονίσω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό και βλέπω ότι στο πρόγραμμά σας δεν του έχετε δώσει μεγάλη σημασία παρόλο που σε αυτή τη χρονική περίοδο οξύνονται οι εξτρεμισμοί, οι ακραίες θέσεις, ο λαϊκισμός, ε, Δηλαδή, ο πολιτισμός μας θα έπρεπε να είναι ο συνδετικός μας κρίκος, είναι, είναι πλούτος και πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και δεν έχετε ε, βάλει την κουλτούρα και τον πολιτισμό ε, ψηλά στις προτεραιότητές σας. Ποια είναι η άποψή σας και για τη διαφοροποιούμενη φορολογία όλων αυτών των κλάδων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα οικοσύστημα με ενιαία φορολόγηση έτσι ώστε ε, να ε, οι επιχειρήσεις όλες αυτές να επωφεληθούν και να φτιάξουν ένα θερμοκήπιο το οποίο θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Και θα μπορούσαμε να ενοποιήσουμε όλα αυτά ή να γίνουν κάποια βήματα. Η Γαλλία έχει τη χαμηλότερη φορολογία, η Ισπανία μέχρι πρώτη την υψηλότερη. Ποια είναι η άποψή σα για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ο κύριος Πόλακ, σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι τονίσατε τις προτεραιότητες της, Φιλανδικής Προεδρίας και δίνετε μεγάλη έμφαση και σημασία στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Ε, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνούμε όλοι στην παραδοχή σύμφωνα με την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην επιτυχία ή μη επιτυχία ενός παιδιού κατά την πορεία του στη συνέχεια στο μέλλον. Έχει φανεί ξεκάθαρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποτυχάνουν στο δικό του σύστημα και όταν με, ταξιδεύουν και πάνε σε κάποια άλλη χώρα τελικά επιτυγχάνουν. Πολλοί φεύγουν από το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και είναι προετοίμαστοι για την αγορά εργασίας. Πώς θα διαδώσετε την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που θα συμπεριλαμβάνει όλους στις πιο μειονεκτικές περιφέρειες της Ευρώπης, σε αυτές που υστερούν περισσότερο, έτσι ώστε παιδιά από δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον να μπορέσουν να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τα καταστήσουν απασχολήσιμα. Ευχαριστώ. Η Υπουργό κυρία Κώσανε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Μπλάνκο για τα ερωτήματά σας. τα οποία είναι όντως πολύ σημαντικά. Ο πολιτισμό, η κουλτούρα στην Ευρώπη είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Ανοίγω λοιπόν αυτό το κεφάλαιο για να πω ότι ε, είναι μια πρωτοβουλία που έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για πολλές πόλεις και περιφέρειες. Η έννοια, για παράδειγμα, της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Είναι και από τις πιο ορατές και εμβληματικές πρωτοβουλίες, άλλωστε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δρούμε σε επίπεδο ατόμων, σε επίπεδο παραγόντων και νομίζω ότι έτσι αναπτύσσεται η, η έννοια της ευρωπαϊκής ε, ταυτότητας και πολιτισμού. Είναι κάτι το καλό. Θα το συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, για τη φορολογία, αυτό είναι αρμοδιότητα Υπουργών Οικονομικών. Κατεξοχήν και αποκλειστικά. Και ε, εξού και η σημασία της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Τώρα, ευχαριστώ κύριε Πόλακ, λέει κύριε Άντερσον, για τη διασφάλιση ποιότητα για τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και την κινητικότητα από το ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο. Ξέρετε, στη σχολική εκπαίδευση, για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διασφάλιση ποιότητα είναι ένα νέο τομέα πάνω στον οποίο θα υπάρξουν συνεργασίε. Πολύ πρόσφατα προέκυψε αυτό ω πεδίο συνεργασιών και ε, άλλωστε το, το, το κράτος διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εμπειροχνωμόνων ειδικών και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανεξάρτητες ερευνητικές αρχές, αν θέλετε, που θα συνεργάζονται με τα εκπαιδευτικά συστήματα για να διασφαλίζουν την ποιότητα, να γίνεται έρευνα για το τι λειτουργεί και το τι δεν λειτουργεί. Και όλα αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν τη διεθνή μας συνεργασία. Άλλος τομέας σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ο δάσκαλος. Βλέπετε ότι εάν υπάρχει υψηλή εκτίμηση στο επάγγελμα του δασκάλου, αυτό ισχύει στη Φιλανδία, και η επαρκής αμοιβή αυτού του επαγγέλματος, ε, αυτά είναι καθοριστικοί παράγοντες για την, ε, την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι έχουν και μεγάλη αυτονομία οι δάσκαλοι ως το περιβάλλον εργασίας, τις συνήθειες εργασίας, τις εκπαιδευτικές και διδακτικές μεθόδους που ακολουθούν και εφαρμόζουν στις διάφορες σχολικές αίθουσες βασικές προτεραιότητες της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και Παιδείας μέχρι το 2025 είναι η άρση των εμποδίων, των φραγμών, το να μπορεί κανείς να σπουδάσει σε ένα άλλο κράτος μέλος, να ενισχύσουμε τη φοιτητική κινητικότητα. Και ε, βλέπουμε ότι σε αυτό υπάρχει πλήρη στήριξη από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και θα περάσουμε τώρα στη τελευταία ομάδα των ε, ερωτήσεων. Σας παρακαλώ τηρήσετε το χρόνο ομιλίας. Ένα λεπτό. Julie Ward, Κολάχα. Ευχαριστώ πολύ. First of all, I'd like to concentrate. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να επικεντρωθώ στο θέμα της κινητικότητας, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι χρησιμοποιώ τον όρο πλέον ε, ελεύθερη κυκλοφορία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως όταν κανείς δουλεύει ε, με ε, παιδιά και με, ε, έχει να κάνει με καλλιτεχνική παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι πολύ σημαντικό για την, τον κλάδο των δημιουργικών να έχει ελεύθερη κυκλοφορία και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ενισχύσουμε. Τώρα όσον αφορά την διαβίου μάθηση και την επικεντρώσή σας, θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, θα εάν ε, θέλετε να κάνετε περισσότερα πράγματα ε, για να προωθήσετε λοιπόν την εκπαίδευση στον τομέα αυτό και όσον αφορά την συμπερίληψη νομίζω ότι το Erasmus συν βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά παραδείγματα επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο άτομα με αναπηρίες ε, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη και που ανέκτησαν έτσι την αξιοπρέπειά τους. Έχω μια... Ε, κάτι τελευταίο να πω. Ε, συνέταξα μια έκθεση για τον πολιτιστικό διάλογο και τις ε, θεμελιώδεις αξίες, ε, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι στην Επιτροπή και για την δήλωση του Παρισιού. Όλοι οι υπουργοί έκαναν λοιπόν μια κοινή δήλωση και θα ήθελα να μάθω αν θα την ακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο υπουργούς για την εξαίρετη παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας. Αναγνωρίζετε ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας ε, είναι κινητήριος δύναμη για όλους τους τομείς και ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το δυναμικό και στον τομέα της παιδείας. Αναγνωρίζεται, λοιπόν τις θετικέ επιπτώσεις τη ψηφιοποίηση στην οικονομία. Παράλληλα όμως, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει και ένας ισχυρός δεσμός με την πρόσβαση στην παιδεία και με την ευημερία. Και ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ναι, στην οικονομική ανάπτυξη τομέα, του τομέα αυτού, αλλά και της ανταλλαγής γνώσεων. Έχετε σχέδια λοιπόν ε, ε, προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της Προεδρίας σας. Ολοκληρώνοντας, κυρία Πιντσουμέα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις δύο Υπουργούς για την παρουσίασή τους. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και διαβάζοντας και τις προτεραιότητες της ε, Φιλανδικής Προεδρίας, αυτό που με ανησυχεί είναι το εξής. Σε ποιο βαθμό σας ενδιαφέρει να καλλιεργήσετε την οτροπία του επιχειρηματία στους νέους, την ε, αίσθηση και την επιθυμία του επιχειρήν, γιατί οι επιχειρηματίες που ε, αναλαμβάνουν ρίσκα, που επενδύουν, που τολμούν, είναι αυτοί που δημιουργούν δημιουργούν πλούτο, που δημιουργούν ανάπτυξη και δίνουν δουλειέ και δημιουργούν απασχόληση. Πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτό το πνεύμα στου νέου, να, να του δώσουμε καλύτερε και περισσότερε δεξιότητε και να έχουν καλύτερη και περισσότερη κινητικότητα. Δουλεύουμε έτσι ώστε τα παιδιά ε, να επιστρέψουν κάποια μέρα από το σχολείο και να πούν στους γονείς τους «Μπαμπά, μαμά, θέλω να γίνω επιχειρηματίας όταν μεγαλώσω». Γιατί αυτό χρειαζόμαστε, ότι είναι καλό πράγμα να καλλιεργήσουμε αυτή την αίσθηση, αυτή την νοοτροπία και να μπορέσουμε να ε, ε, κάνουμε αυτή την εκπαίδευση για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να ανοίξουν οι δουλειές. Ευχαριστώ. Um, thank you, Mrs. Ward, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βόρτ, και τους άλλους δύο που έθεσαν ερωτήσεις. Ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχήν το θέμα της διαβίου κατάρτισης, της συνεχούς κατάρτισης και της ψηφιοποίησης. Βεβαίως εδώ πολλά συμπληρωματικά βήματα πρέπει να γίνουν για να ενισχύσουμε αυτήν την διαβίου κατάρτιση, μάθηση η έννοια της ε, συνεχούς μάθησης βεβαίως αφορά άμεσα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά της εργασίας και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς ανταποκρίνονται ατομικά αυτοί που θέλουν διαρκώς να αποκτήσουν νέα προσόντα και να βελτιώσουν ε, τις δεξιότητές τους, αλλά και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Χρειαζόμαστε πιο μεγάλη ευελιξία, πιο ευέλικτα συστήματα και κυρία Ward έχετε δίκιο, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και στις ανάγκες των εργαζομένων. Όταν μιλάμε για ενήλικες οι οποίοι θέλουν να ενσωματωθούν σε αυτήν την διαδικασία διαρκούς κατάρτισης και συνεχούς μάθησης, ε, συνήθως προσκρούμε σε δυσκολίες που αφορούν κυρίως έλλειψη χρόνου, έλλειψη χρημάτων, κάτι που τελικά τους αποθαρρύνει. Σας ευχαριστώ όλους πάντως για τις ερωτήσεις σας για την έμφαση που δίνεται στις αξίες, στις αξίες ευρωπαϊκές, στις κοινωνικές αξίες και στο πώς η πολιτική μας μπορεί να τη στηρίξει. Ολοκληρώνω με την τελευταία ερώτηση. Νέοι επιχειρηματίες, επιχειρηματικότητα των νέων. Αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Πώς δηλαδή δίνουμε τα εργαλεία σε αυτούς τους νέους, οι οποίοι το επιθυμούν, να γίνουν επιχειρηματίες. άμεση σχέση έχει με το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόσονεν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Κυρία Ward, το Συμβούλιο θέλει να στηρίξει την κινητικότητα στα πλαίσια της Δημιουργικής Ευρώπης, της πρωτοβουλίας αυτής. Οι γνώσεις, η καινοτομία είναι καθοριστικές για την πρωτοβουλία αυτή. Την ίδια ώρα όμως θέλουμε να επιμείνουμε σε θέματα που αφορούν την ισότητα, την κατάρτιση, τη βιωσιμότητα αυτών των δράσεων. Η Ατζέντα 2030 είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Είναι στόχος τον οποίο μοιραζόμαστε και θεωρούμε ότι ο πολιτισμός φυσικά ε, ενσωματώνεται στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και δεν μας ενδιαφέρει μόνο να στοχεύσουμε στον πολιτισμό και σε πολιτιστικούς μόνο στόχους. Έχουμε και πολλά άλλα στοιχεία και προγράμματα τα οποία εμπεριέχουν μία πολιτισμική συνιστόσα. Επίσης, σε όλους τους πολιτικούς τομείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο πολιτισμός είναι καθοριστικός για την ενίσχυση της δημοκρατίας, είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν δυνατή πολιτική στον τομέα του πολιτισμού. Χρειαζόμαστε αποφασιστικές δράσεις. Το Συμβούλιο λοιπόν θα παίξει καθοριστικό ρόλο εδώ, γιατί το Συμβούλιο αποφασίζει. Θα δούμε βέβαια τι θα προτείνει και η νέα Επιτροπή στον κοινωνικό τομέα. Αυτό που είναι σημαντικό όλοι μαζί να συμφωνήσουμε ότι αυτός ο πολιτισμός, αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη και η πολιτιστική συνιστόσα της αποτελούν τον καθοριστικό άξονα δράσης για μας. Μιλήσατε επίσης για την επιχειρηματικότητα των νέων. Θέσεις απασχόλησης, ποιοτικές θέσεις, για τους νέους είναι προς όφελος της απασχόλησης, αλλά είναι κυρίως προς όφελος των νέων και της ενσωμάτωσης τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ την κυρία Άντερσεν, ευχαριστώ την κυρία Κόσονεν. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ εντατική συνεργασία και τους επόμενους τέσσερις μήνες της Φιλανδικής Προεδρίας. Σίγουρα ο τριμερής διάλογος θα ξεκινήσει, όπως μας είπατε, σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you. It was really very interesting and yeah. I think good hearing. Okay. Thanks a lot. Thanks. Thanks.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

Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο Γενικός Διευθυντής της DG Connect θα μας κάνει μια παρουσίαση, ο Ρομπέρτο Βιόλα. Σας παρακαλώ πολύ, όποιος θέλει να βγει μπορεί να το κάνει με συντομία και σιωπηλά παρακαλώ tightly and fast, because we have still points on our agenda. And I want to ask the colleagues to take their seat. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Καθίστε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την συνεδρίασή μας. Ja, ich Όπως μόλις σας είπα, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Ρομπέρτο Βιόλα, Γενικό Διευθυντή της DG Connect. Είναι μεγάλη χαρά για μένα κύριε Βιόλα που σήμερα σας έχουμε εδώ μαζί μας στην Επιτροπή. Θα συζητήσουμε μια σειρά πολύ ενδιαφέροντων θεμάτων και σημείων. Το θέμα των ψευδών ε, ειδήσεων, παραδείγματος χάρη είναι κάτι που έχει απασχολήσει την Επιτροπή και εμάς, η ουδετερότητα των δικτύων, του διαδικτύου, το θέμα της α, υπηρεσίας 5G. Αναφέρθηκα απλώς σε κάποια από τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μας. Το θέμα Euronews επίσης, το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει κάποιους από τους συναδέλφους, ήδη το θίξαμε. Έχετε για 10 λεπτά το λόγο, κάντε μας μια σύντομη παρουσίαση και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και η συζήτηση. Κύριε Βιόλα, έχετε το λόγο. Dear Madam Chair, honorable members of the committee, Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη της, Ευρω... Ε, της Επιτροπής σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είναι και τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να σας παρουσιάσω την δουλειά η οποία γίνεται προκειμένου να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη θητεία της. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι Έχουμε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές από την εκλεγήσα ε, πρόεδρο Μιλούμε για την ψηφιακή μετάβαση. Μιλούμε για το μέλλον της Ευρώπης. και όλοι οι τομείς που μας απασχολούν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την Πρόεδρο και θα περιμένουμε ε, την ε, ανάθεση των χαρτοφυλακίων στους επιτρόπους, τις ακροάσεις τους και την ε, πλήρη δρομολόγηση και εύρυθμη κανονικότητα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα νομοθετικά καθήκοντα που πρέπει να ασκήσουμε και ήδη είμαστε πολύ απασχολημένοι και προσπαθούμε να τα εκπληρώσουμε σωστά. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. θα κάνουμε δουλειά για την ε, οδηγία για το Media Service. Εδώ και τρία χρόνια έχουμε εργαστεί επισταμένος. Ε, ταξίδεψα παντού στον κόσμο και συνειδητοποίησα ότι εμείς είμαστε η πιο προχωρημένη σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύγκληση των παραδοσιακών ΜΜΕ, των κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως είναι το Video On Demand και το καθεξής. Δηλαδή η σύγκληση στην Ευρώπη μεταξύ όλων αυτών είναι μεγαλύτερη από όπου, οπουδήποτε αλλού. Και πρέπει να δούμε το θέμα της διανομής, περιεχ... όποια μορφή και αν πάρει αυτό το περιεχόμενο. Επομένως, νέο χαρακτηριστικό της οδηγία αυτής είναι ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο video sharing platform. Έχουμε έμφαση έμφαση στο παιχνίδι επί ίσης όρους, οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν με τα, ε, στα παραδοσιακά μέσα και στο video on demand και στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοντολογία, με, την, ε, με το διοκτησιακό καθεστώς, με την προστασία των ανηλίκων, οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Και Από την έγκριση της οδηγίας ε, και μετά, εάν χρειαστεί περισσότερη ε, διευκρίνηση, θα το κάνουμε για να προστατεύσουμε τους πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο για για το βίντεο για το Christchurch και όλα αυτά έδειξαν ε, ανέδειξαν την ανάγκη αυτή και καλύπτεται στην οδηγία για το media service. Άρα θα είναι οδηγία πρότυπο. Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της οδηγίας αυτής είναι ότι για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών των ε, οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να έχουμε πλουραλισμό θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη τοπική ρυθμιστική αρχή, ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Θα είναι νομική παράμετρος αυτή για να κρίνουμε την ανεξαρτησία συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Άλλωστε, πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά είναι η συνεργασία των νομοθετών. Το έργα είναι μια ομάδα Ευρωπαίων νομοθετών και αποτελεί μέρος της οδηγίας. Έχει συσταθεί επισήμως. Είναι ένας νέος μηχανισμός, καινούριο, εξαιρετικά σημαντικός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να παρακολουθήσουμε την ενσωμάτωση όλων αυτών στην εθνική νομοθεσία με καταληκτική προθεσμία το Σεπτέμβριο του 2020 και θα ασκήσουμε επίσης στα κράτη-μέλη για να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και αυτό το οποίο θα κάνουμε επίσης είναι να διευκολύνουμε την ε, εφαρμογή, την υλοποίηση της οδηγίας. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές κυρίως για τα μέσα κοινωνική δικτύωσης και για τα κριτήρια για την απαραίτητη λειτουργικότητά τους τα μέσα κοινωνική δικτύωση ε, αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας και η οδηγία λέει ότι όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση που έχουν το βίντεο ω απαραίτητη λειτουργικότητά τους θα υπάγονται στην οδηγία. Άπαξ και ενσωματώνουν βίντεο ω απαραίτητη λειτουργία και θα διαμορφώσουμε και θα διατυπώσουμε αυτά τα κριτήρια με τρόπο κατά τον οποίο να παράγουν νομικό αποτέλεσμα και να οδηγούν στην ταυτοποίηση αυτών των πλατφορμών και την αναγνώριση αυτών με το, όσο τον πιο ομοιόμορφο τρόπο. Το θέμα του 30% και της ποσόστοσης, το οποίο απαιτείται από οποιοδήποτε πάροχο video on demand, πλατφόρμες όπως το Netflix, πρέπει να συμμορφωθούν με την οδηγία και το 30% του περιεχομένου τους να είναι ευρωπαϊκό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κριτήρια μας είναι απλά, είναι εύκολα, είναι σαφή και οδηγούν στην ομοιόμορφη ερμηνεία της ε, οδηγίας στο βέλτιστο δυνατό βαθμό. Άλλο στοιχείο της οδηγίας θα είναι και η εξαίρεση. Λέει η οδηγία ότι επαλλάσσονται οι μικρές επιχειρήσεις. Πώς προσμετρώνται όμως, πώς υπολογίζονται ως μικρές αυτό θα διαμορφωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές. Άρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα, εκπονούμε ένα προσχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσουμε στα κράτη-μέλη, θα γίνει αντικείμενο συζήτησης, θα ξεκινήσει η συζήτηση επ' αυτού. Και, και θα το διαθέσουμε Έχουμε ένα κώδικα δεοντολογία, τον οποίο προσυπογράφουν όλο και περισσότερε επιχειρήσει. Και τώρα, μετά τι ευρωπαϊκέ ορίζοντα 2020 και θα ε, κάνουμε ένα διαγωνισμό για ύψους ύψους ε, ευρώ. Θέλουμε δηλαδή να προχωρήσουμε ε, με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πρόγραμμα και θα έχουμε περισσότερα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση και προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα προγράμματα πολιτισμού και για το ευρύτερο πλαίσιο για τον πολιτισμό. 75 εκατομμύρια ευρώ θα είναι αυτά που θα δοθούν για τα οριζόντια ζητήματα για όλα τα μέσα. Βεβαίως όταν μιλούμε για πολιτιστικά προγράμματα εννοούμε το Creative Europe. Δεν το είπα ξεκάθαρα, αλλά είναι σαφέ. Άλλωστε, σε λίγε μέρες θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Για το Creative Europe το σημαντικό είναι ότι ο επιτρόπο ζήτησε 30% αύξηση του προϋπολογισμού και το Κοινοβούλιο αποφάσισε να πάει ακόμη πιο πέρα. Σε κάθε περίπτωση είναι 0,01% του προτινόμενου προϋπολογισμού. Τι πιστεύετε, αξίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμό περισσότερα ή αξίζει μόνο το 0,01% του προπολογισμού μας. Είναι δυσάρεστο το καθήκον για το Συμβούλιο να περικόψει ή το Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή να περικόψει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά οι οριζόντιες μειώσεις στον πολιτισμό είναι πισόπλατη μαχαιριά. Βεβαίως προτείνουμε εμεί αύξηση. Το Κοινοβούλιο προτείνει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, αλλά είναι πολύ λίγο ο προπολογισμό που ε, καλούμαστε να υπερασπιστούμε. Ζητούμε από όλα τα κράτη-μέλη να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία ε, για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ε, τρισδιάστατων εικόνων για τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με, την, ε, ε, με το δραματικό συμβάν της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων επιβεβαιώθηκε αυτή μας η επιθυμία ότι πρέπει να υπάρχουν τρισδιάστατες εικόνες απεικόνησης της ε, πολιτιστική μας κληρονομιάς. Και ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία το γεγονός, το ευτυχές γεγονός ότι υπήρχε αυτή η απεικόνηση για την Παναγία των Παρουσίων. Εμείς όμως θέλουμε αυτό να το πράξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κράτη, ε, και ε, είναι πολύ σημαντικό για όλους. Τώρα για την ουδετερότητα των μέσων, γιατί έχω ξεπεράσει τα 10 λεπτά, έχουμε αξιολογήσει το εξής. Μόνο εμείς έχουμε νομοθεσία για την ουδετερότητα του διαδικτύου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεχάσει ο κόσμος τι συνέβαινε όταν ε, σε άλλες χώρες του κόσμου και σε άλλες περιοχές το Skype είχε μπλοκαριστεί, το WhatsApp ή δεν μπορούσε αυτά να τα κατεβάσει κανείς και να τα χρησιμοποιήσει σε κινητό γιατί θα μπορούσε να μετακινηθεί και να τα χρησιμοποιήσει και από αλλού. Επομένως, ε, ε, όλα αυτά λειτουργούν σωστά στην Ευρώπη. Πολλοί λένε ότι το 5G θα αλλάξει την ε, την κατάσταση. Εμείς δεν το συμμεριζόμαστε αυτό. Πιστεύουμε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ισχύει και για το 5G και θα ταιριάσει μια χαρά. θα πρέπει να υπάρχει ένα μέρος του φάσματος κάτω από τα 700 MHz, το οποίο να δοθεί για το broadcasting. Και αυτή είναι και η δική μας θέση. Ε, όταν το, τα ενέκρινε αυτά ε, το Συμβούλιο τον Ιούνιο στην Παγκόσμια Ραδιοφωνική Διάσκεψη για τα θέματα αυτά ραδιοκυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παραμένει προσιλωμένη στην ιδέα ότι το ραδιοφωνικό φάσμα θα ε, πρέπει να δίδεται και για το broadcasting μέρος αυτού και να υπάρχει εγγύηση από αυτού. Θέλουμε το πρασίνισμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Έχει υποθεί ότι τα, τις πρώτες 100 μέρες θα υπάρξει νομοθεσία για τη τεχνητή νομοσύνη και την περασμένη εβδομάδα στη Βενετία είδαμε ότι πολλοί σεναριογράφοι ήδη σκέπτονται να έχουν προ... χαρακτήρες τεχνητής νομοσύνης στις ε, ταινίες τους. Είναι κάτι που αφορά άμεσα τον τομέα του πολιτισμού. Είναι κάτι που έχει άμεσες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και στον τρόπο ύπαρξής μας ως Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό θα είναι διακλαδική, διατομεακή αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σταματήσω κάπου εδώ. Υπάρχουν και πολλά άλλα, πολλά και ενδιαφέροντα. Ε, με χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις και θα διευκρινίσω οτιδήποτε έχει παραμείνει εκρεμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πινκ-πονγκ. Ερώτηση-απάντηση. Ξεκινήσουμε με τους ε, εισηγητές. Η κυρία Σόντροβα. Σας ευχαριστώ για την ε, πρώτη σας παρουσίαση. Βεβαίως και έχουμε ερωτήσεις που αφορούν τα διάφορα δίκτυα και κανάλια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Η οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και βεβαίως ε, έχουμε ακόμα κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την προώθηση των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε επαφές με τα κράτη-μέλη, έχετε κάπως πιο συγκεκριμένα πάρει θέση και έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δείτε ποιες είναι οι νομοθετικές τους δυνατότητες, πόσο έχουν προετοιμαστεί, και τι ακριβώς έχουν κάνει για την υλοποίηση. Εμείς σαν βουλευτές έχουμε κάθε συμφέρον να συνεργαστούν σωστά τα κράτη-μέλη μας, έτσι ώστε η ερμηνεία και η υλοποίηση αυτών των νέων ε, κανόνων να είναι επιτυχής και αποτελεσματική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα θέλαμε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν και να λειτουργήσει αυτή η νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Βιόλα. Βεβαίως και δίνουμε μεγάλη σημασία σε μια ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή ε, της οδηγίας και παρακολουθούμε στενά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και την εξέλιξη ε, στα κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε όλο αυτό θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2020. Όλοι μιλούν για το HPH, όλοι μιλούν για τα κοινωνικά δίκτυα. Ποια είναι όμως η ευρωπαϊκή νομοθεσία Υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός και η υλοποίηση αυτής της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί με τον πιο ομοιόμορφο δυνατό τρόπο. Έχουμε τις κατευθυντήρες γραμμές, έχουμε την ομάδα επαφής, την παρακολουθούμε και τη συνοδεύουμε στα διάφορα στάδια και βεβαίως ε, θα δούμε πώς μεταφέρονται και πώς μεταφράζονται στην Εθνική Νομοθεσία όλα αυτά. Η κυρία Κάμερφελ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βιόλα. Έχω άπειρες ερωτήσεις. Όσον αφορά την ε, υλοποίηση της οδηγίας, ε, χαίρομαι που το βάλατε σαν κεντρικό σημείο της παρουσίασή σας. Μιλήσατε για απλό και εύκολο περιγράφοντας τη διαδικασία υλοποίησής της και εφαρμογής της. Εγώ όμως βλέπω στην πράξη το αντίθετο. Δηλαδή μόνο 30% ευρωπαϊκών ε, έργων και δημιουργημάτων βλέπουμε να βρίσκονται στις πλατφόρμες μέχρι τώρα. Αυτό το 30% αν θέλουμε να το διατηρήσουμε, είναι τελείως παράλογο. Σαν νομοθέτης πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και στην πράξη να μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό το περιεχόμενο το ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκής προέλευσης, να το εξασφαλίσουμε και να μην υπάρχει απολύτως καμία αβεβαιότητα. Όσον αφορά το άρθρο 13, loading και loading over πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Στην πράξη μου φαίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας SNCL, το περιεχόμενο το οπτικοακουστικό στις πλατφόρμες, το θέμα της, του πόσο δημοφιλής είναι μια υπηρεσία, μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Εάν θέλουμε να κρατήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας, θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς θα δώσουμε δυνατότητε σε όλες αυτές τις πλατφόρμες να διοχετεύουν με αποτελεσματικό τρόπο όλα αυτά τα ευρωπαϊκά δημιουργήματα, το ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Αλλιώς πραγματικά δεν χρειαζόμαστε αυτά τα κριτήρια. Υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα, λειτουργούν και κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσει η Επιτροπή σε σχέση με τις προτάσεις του Συμβουλίου μέχρι το 2030 όσον αφορά το, τις συχνότητες και τα 7 MHz. Εδώ χρειάζονται τεχνολογικές εξελίξεις που θα προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση. Θα σταματήσω εδώ γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, τις οποίες αν μου δοθεί ευκαιρία θα τις κάνω λίγο αργότερα. Κύριε Βιόλα, έχω και εγώ μια άμεση ερώτηση που να σας κάνω όσον αφορά τις συχνότητες, τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Αυτό το εύρος συχνοτήτων και τα 700 παραδείγματο χάρη αφορά μόνο το ραδιόφωνο, γιατί τι ακριβώς θα γίνει με το θέατρο και με άλλους τομείς. Θα ανανεωθούν, αν θέλετε, με την απελευθέρωση των συχνοτήτων και αυτοί οι τομείς. Έχετε συμπεριλάβει στην πολιτική σας την προοπτική επενδύσεων και σε θέατρα, αλλά και σε άλλους τομείς της ψυχαγωγίας και της δημιουργίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάμερβερ, αναφέρθηκε στις κατευθυντήρες γραμμές. Καταρχήν, ναι, όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Το επεξεργαζόμαστε και εσείς αναφερθήκατε στο δύσκολο σημείο. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι το ένα θέμα που μπορούμε εμείς να προετοιμάσουμε. Απ' την άλλη είναι πώς θα μεταφερθούν αυτά στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Και ο μόνος τρόπος να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη και σοφή λύση είναι να ακούσουμε προσεκτικά τις απόψεις όλων μέχρι να φτάσουμε στην πιο ικανοποιητική λύση. Μιλήσατε επίσης και για ένα άλλο επίμαχο σημείο, το 30%. Κοιτάξτε, βεβαίως εδώ υπάρχουν σειρές οι οποίες μπορεί να καταναλώσουν πολύ γρήγορα αυτό το 30%. Καταλαβαίνετε όμως ότι μία σειρά είναι ένα μια κινηματογραφική ταινία η οποία ε, ουσιαστικά παρουσιάζεται σε πολλά επεισόδια, μια μακρύτερη ε, κινηματογραφική ταινία. Πώς λοιπόν θα καλύψουμε τους ε, υπάρχοντες ορισμούς χωρίς να εξαντλήσουμε αυτό το 30%. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αχαρτογράφικα νερά. Είναι κάτι το εντελώς καινούριο. Καταλαβαίνω τι λέτε, Και βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το κείμενο της οδηγίας. Μιλάει για δημοφιλή περιεχόμενο. Δημοφιλές περιεχόμενο, συγγνώμη. Ε, μα δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι είναι δημοφιλές, ότι θα είναι και αυτό το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε σαν ουσιαστικό περιεχόμενο. Κοιτάξτε, παραδείγματος, χάρη τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα και την έκφραση της υποστήριξης με τα likes. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να το δούμε αυτό σαν ένα συμπληρωματικό στοιχείο. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στην φάση ολοκλήρωσης του σχεδίου. Η ομάδα επαφής, οι, οι και οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων θα συνεχίσουν τις συζητήσεις. Είμαστε δε εντελώς ε, στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να έρθουμε και να σας παρουσιάσουμε τα επόμενα βήματα της διαδικασίας όσον αφορά την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών. Επίσης μιλήσατε και για τις συχνότητες. Είναι σαφές ότι η απόφαση για τα 700 MHz και για τα σύρματα μικρόφωνα επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό. Είναι απόφαση της Επιτροπής και πιστεύω ότι οι λύσεις που έχουμε βρει είναι ικανοποιητικέ. Βεβαίως, όσον αφορά τα σύρματα μικρόφωνα, θα πρέπει να εντοπιστούν και άλλες λύσεις και εδώ είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φερό. Merci, Monsieur le Directeur Général. Ευχαριστώ κυρία Γενική, Γενική Διευθυντά. Δεν γνώριζα αυτή την πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και σας συγχαίρω. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια, ποιο είναι το θεματολόγιο, ε, αν, υπάρχει, αν έχει ξεκινήσει κάτι ήδη. Και μια άλλη ερώτηση. που έχει να κάνει με το ρυθμιστικό κομμάτι το οποίο εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο όσον αφορά την παιδεία και το επιγραμμικό περιεχόμενο. Υπάρχει αυτή η οδηγία και η οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα ε, την οποία υποστηρίξαμε και το δίκτυο λοιπόν για την δορυφορική τηλεόραση. Η τεχνολογία λοιπόν εξελίσσεται συνέχεια, είναι πολύ σημαντικό να προσαρμόσουμε το νομοθετικό μας πλαίσιο ε, και να μεριμνήσουμε για τον ψηφιακό τομέα. Όσον αφορά αυτό το 30% την ποσόστοση για τα ευρωπαϊκά έργα, νομίζω ότι δεν εφαρμόζεται σήμερα στις μουσικές πλατφόρμες και είναι ένα πραγματικό πρόβλημα αυτό. Διότι ε, αυτό έχει να κάνει και με τα βίντεο αλλά έχει να κάνει και ε, με τους αναζητητές ε, στο ίντερνετ. Όπως ε, για παράδειγμα όταν ψάχνετε κάτι στο YouTube, δεν υπάρχει εδώ λοιπόν μία αντιστοιχία με αυτή την θέληση προώθησης του ευρωπαϊκού περιεχομένου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρύθμιση για το επιγραμμικό περιεχόμενο και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού περιεχομένου, η σωστή αμοιβή των δημιουργών και ε, να κάνουμε πιο υπεύθυνες τις πλατφόρμες. Ε, ο ψηφιακός τομέας μένει ένας χώρος δημοκρατίας και παραμένει ένα τεράστιο διακύβευμα του μέλλοντος. Οι νομοθέτες λοιπόν δεν θα πρέπει να ε, αφήσουν να τους ξεπεράσει η καινοτομία. Εμείς έχουμε φόβους επ' αυτού. Πώς λοιπόν ε, η Κομισιόν θα παρακολουθήσει την εφαρμογή της οδηγίας που συζήτησαμε πριν από λίγο, την γρήγορη εφαρμογή της. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει ήδη μια νομοθεσία ε, όσον αφορά το επιγραμμικό και μη περιεχόμενο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν για την εφαρμογή και το επόμενο διακύβευμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η πολύ γρήγορη ανάπτυξη, ίσως πιο γρήγορη από την ικανότητά μας να νομοθετούμε, οι τεχνολογικές εξελίξεις. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να κάνουμε όλο αυτό το έργο και πώς θα μπορέσουμε να το προσαρμόζουμε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, την ψηφιοποίηση δηλαδή της, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και το πρόγραμμα για το οποίο σας μιλήσαμε, έχουμε, είχαμε το πρόγραμμα Europeana και συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτή την βάση δεδομένων για ψηφιοποίηση των έργων πολιτισμού. Θα ε, δούμε και με την UNESCO πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια και να της δώσουμε ε, νέες προοπτικές. Ξεκινήσαμε ήδη με μια ομάδα τεχνική σε επίπεδο κρατών μελών και περιμένουμε ανυπόμονα επίσης ε, χρηματοδότηση από το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αυτό θα ενταχθεί στο πρόγραμμα για, και την χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το σύνολο νομοθετημάτων που εγκρίθηκαν κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο. Ε, ήταν αρκετά εντυπωσιακά όλα αυτά, ε, γιατί ε, όπως είπατε μιλούσαν για το copyright, για τα πνευματικά δικαιώματα και είχαμε και τους ε, κανόνες για την ε, τηλεπικοινωνία. Και όλα αυτά ε, αφορούσαν όλα τα κράτη-μέλη. Ήταν κάτι επίγον να έχουμε μία συνεκτική και μία καλή εφαρμογή. Υπάρχει όμως το τεχνικό πρόβλημα ότι όσον αφορά την δορυφορική τηλεόραση, όσον αφορά το copyright, όλα αυτά θα εφαρμοστούν μετά από κάποια άλλα πράγματα που έχουν αποφασιστεί πριν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική θεώρηση όλων αυτών. Όσον αφορά το copyright, εμείς ε, θέλουμε να κάνουμε έναν ε, διακρατικό διάλογο για την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας. Κάναμε λοιπόν μια έκκληση ούτω ώστε να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος πάνω στο άρθρο 17. Και βεβαίω έχουμε καταβάλει πολλέ προσπάθειες για να παρέχουμε συνδρομή στα κράτη-μέλη. Και όπως είπα και πριν, ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν θα αρχίσουν να κάνουν το καθένα δική του νομοθεσία, αλλά θα παραμείνουν στον κύριο δρόμο. Δηλαδή, να εφαρμόσουν το σύνολο όλες αυτές τις οδηγίες, ούτω ώστε να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Όσον αφορά την ποσόστοση 30%. Ναι, αναφέρεται στα οπτικοακουστικά μέσα. αλλά όσον αφορά τις πλατφόρμες Video On Demand θα δοθεί ε, εκεί προτεραιότητα. Και αυτό εφαρμόζεται και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες που προσφέρουν ε, βίντεο επιπληρωμή ή όχι. Και σε αυτή την ε, περίπτωση λοιπόν θα ισχύουν τα κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βιόλα για τα σχόλιά σας. Με θετικό μάτι βλέπω την ε, επιθυμία σας να παρακολουθήσετε περισσότερο την παρουσία των ευρωπαϊκών έργων τα κοινωνικά μέσα και στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Με ποια μεθοδολογία όμως και όταν ε, αποκτήσετε αυτά τα δεδομένα, τι θα κάνετε με αυτά. Και αν ε, τα δεδομένα σας, λένε ότι δεν τηρείται αυτή η ποσόστοση, τι θα κάνετε. Και για την πληροφόρηση, αν κατάλαβα καλά, περισσότερα κονδύλια προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά. Μας λέτε πιο συγκεκριμένα ποιες δράσεις θα στηριχθούν. Έχετε προοδεύσει στο διάλογο που κάνετε με τους βασικούς παίκτες όπως είναι το Facebook. Είναι δύσκολη η συνεργασία με αυτούς αλλά χωρίς συνεργασία με αυτούς δύσκολα θα καταφέρετε κάτι στις πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος για τα ηθικά ζητήματα, για τη τεχνητή νοημοσύνη, τι θα κάνετε. Θα θετήσετε μέτρα για τον περιορισμό και τον αποκλεισμό των εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να χειραγωγήσουν τη συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου. Ευχαριστώ πολύ. Για την ποσόστοση του 30% Εάν μια πλατφόρμα ή ένα βίντεο on demand δεν τηρεί το 30% θα παραβαίνει την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Και βασικός ρόλος ε, παίζεται από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή η οποία θα πρέπει να ελέγχει και η οποία θα πρέπει να συμφωνήσει για τα κριτήρια ελέγχου με τις λοιπές ρυθμιστικές αρχές της κατατόπους ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός θα είναι ο βασικός μηχανισμός ελέγχου. Θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία, ύπαρξη του αριθμού των έργων στις πλατφόρμες, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα αποθετήριο ε, των ευρωπαϊκών έργων η ιδέα ενός index είναι πιο απλή. Να τα μετρήσει κανείς άπαξ και τα έχει εντοπίσει, τα έχει αναγνωρίσει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καταλογοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά έργα και θα κάνουμε μια μεγάλη δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Τώρα από πλευράς δραστηριοτήτων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους διακριβωτές γεγονότων, τους fact-checkers, για να συνεργάζονται. Δεν θα τους χρηματοδοτήσουμε γιατί έτσι θα ήταν σαν να φτιάχταμε ένα Υπουργείο Αλήθειας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουν ένα ασφαλή χώρο, γιατί έχουν υποστεί ε, ε κυβερνοεπιθέσεις στο παρελθόν, ότι ε, έχουν ένα ασφαλή χώρο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες, για να συνεργάζονται, να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος της ομάδας μας. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία των μεγάλων πλατφορμών, σαφέστατα προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό θεωρούμε ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι έχουν αυτοδεσμευτεί σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την έκκληση για αυτορύθμιση. Και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούν και θα καταλάβουν ότι, το ότι η οδηγία αυτή είναι κάτι το πολύ σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει την άλλη κληρονομιά και το περιεχόμενο στις πλατφόρμες. Όταν η πρόεδρο ανακοίνωσε την ύπαρξη νομοθεσία για την τεχνητή νομοσύνη τι πρώτε 100 μέρε τη θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί με ευρωπαϊκό τρόπο αυτή η νομοθεσία, ε, ήξερε πολύ καλά και εμεί συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με ε, τους αρμοδίους πρέπει να επιβάλλουμε ε, και να διατυπώσουμε οι κώδικα διοντολογίες, ηθικές κατευθυντήριες γραμμές και σε θελούσια βάση ήδη τις εφαρμόζουν ορισμένες επιχειρήσεις. Στα τέλη της χρονιάς θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα ε, ως προς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέω ο κύριος Νίνας. Οι ερωτήσεις που έκανε εκεί η κυρία Κάμερβερτ αλλά και άλλοι με βρίσκουν ε, σύμφωνο. Όσον αφορά τώρα τα τρισδιάστατα μοντέλα, την τρισδιάστατη αποτύπωση, μπορείτε να μας ε, δώσετε κάποια στοιχεία όσον αφορά τον τομέα αυτό. Μίλησατε επίσης για το 30% αύξηση για το πρόγραμμα Creative Europe. Εμείς ε, πολύ θα θέλαμε. Αυτό είναι μία απέτηση, θα έλεγα, της δικής μου γενιάς, των νέων της Ευρώπης, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε πραγματικά μια ευρωπαϊκή ταυτότητα στον πολιτιστικό τομέα και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε πραγματικά την ε, ευρωπαϊκή δημιουργικότητα. Επίσης, οι πλατφόρμες. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το περιεχόμενο. Και εδώ εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα της χρηματοδότησης και του κόστους. Να έχουμε δηλαδή καλύτερες επιλογές όσον αφορά το τι ευρωπαϊκό περιεχόμενο ε, αγοράζουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί από τη φάση της επιλογής, γιατί το κόστος βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, είναι πολύ πιο χαμηλό αλλού εκτός Ευρώπης. Το θέμα όμως δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό το κριτήριο. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, υπάρχουν προσπάθειες από μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί το δημιουργικό κομμάτι και ιδιαίτερα στην ε, βιομηχανία του κινηματογράφου. Σήμερα υπάρχουν ε, τεράστια προβλήματα όσον αφορά και ε, το ψηφιακό περιεχόμενο. Ποια είναι λοιπόν η προσπάθεια της Επιτροπής και όσον αφορά τον προγραμματισμό και όσον αφορά την παραγωγή και όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των ε, κινηματογραφικών ε, και άλλων ε, δημιουργημάτων τα οποία πραγματικά σαν έργα πολλές φορές θέλουμε να στηρίξουμε. Το Spotify, αλλά όχι μόνο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουν αυτό το ποσοστό ευρωπαϊκό περιεχομένου. Ποιος κάνει την επιτήρηση, ποιος κάνει τον έλεγχο. Και ολοκληρώνοντας για το Euronews θα ήθελα να ρωτήσω τι έχετε να πείτε για τη χρηματοδότησή του και για τις ψευδείς ειδήσει, το fake news, τι έχουμε σήμερα, τι δυνατότητες έχουμε σήμερα να επαληθεύσουμε το περιεχόμενο και την αλήθεια κάποιων πληροφοριών, ιδιαίτερα στο deep fake. Πρόεδρος, πολλές ερωτήσεις, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ναι, θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα και με συντομία. πάρα πολλές και πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Όσον αφορά τα μοντέλα τα τρισδιάστατα, το θέμα δεν είναι απλώς αυτά να είναι διαθέσιμα για να προστατεύσουμε αυτήν την δυνατότητα, την τεχνολογική, αλλά και τη δημιουργικότητα, αλλά να βασιστούμε και εδώ στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία εδώ να χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτήν την νέα ανάγκη για να δημιουργήσουμε νέες ευρωπαϊκές δυνατότητες. Για τους δημιουργούς. Υπάρχει σήμερα αυτή η οδηγία, αυτή η αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρξει μία δίκαιη και αξιοπρεπής αποζημίωση για τους Ευρωπαίους δημιουργούς. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά έργα να προστατεύονται και να ανταμείβονται. Μιλήσατε για την αύξηση της χρηματοδότησης σε όλα τα προγράμματα που αφορούν τα μίντια και ιδιαίτερα για το μίντια. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι γιατί τελικά βλέπουμε ότι οι πιο πολλές ε, δημιουργίες που στηρίχτηκαν δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλουμε περισσότερη λοιπόν ευρωπαϊκή δημιουργία, αλλά θέλουμε περισσότεροι Ευρωπαίοι να ενδιαφέρονται για αυτά τα έργα που στηρίζουμε και που δημιουργούνται. Είναι και το θέμα βεβαίως της δημοσιοποίησης, της επικοινωνίας, της διανομής. Σήμερα μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, των ευρωπαίων δημιουργών, προωθούνται και είναι εύκολο να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Πολλές φορές είναι πιο εύκολο να βρει κάποιο ένα ευρωπαϊκό έργο σε μια αμερικανική πλατφόρμα από ό,τι στις δικές μας. Είναι λοιπόν και θέμα διανομής και θέμα επικοινωνίας και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Μιλήσατε επίσης και για το θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου της χρηματοδότησης κάποιων τομέων όπως το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της χρηματοδότησης ε, του Euronews. Ναι, εμείς βεβαίως στην αποστολή μας, στην εντολή μας, είχαμε την εξέταση του θέματος αυτού. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, η νέα οδηγία. Θα περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η νέα κατεύθυνση στην οποία θα οδηγηθεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, θίξατε και το θέμα του deepfake των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο. Ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, ο μοναδικός σκοπός αυτών των ειδήσεων είναι να αποσταθεροποιήσουν την κοινή γνώμη τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι αρμόδιοι για την επαλήθευση αυτών των ειδήσεων χρησιμοποιούν όλες τις τεχνολογίες και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανταποκριθούν σε αυτό το δύσκολο έργο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Πέζερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενική Διευθυντή, που ήρθατε σήμερα εδώ, σε αυτήν την Επιτροπή. Το πρώτο μου ερώτημα πληροφορήθηκα, μπορείτε να μου πείτε αν είναι έτσι ή όχι, ότι αλλάζεται διατύπωση. Δηλαδή, αντί να μιλάτε πλέον για πολιτιστικό κλάδο, μιλάτε για ε, κλάδο περιεχομένου. Είναι αλήθεια και ποιοι είναι οι λόγοι, εάν αυτό ισχύει. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι όσον αφορά λοιπόν τον κλάδο της δημιουργίας, θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την ε, κοινωνία και την καινοτομία, να υπάρχει ένας ισχυρότερος δεσμός ανάμεσά τους ε, και να μπορέσουμε να στηρίξουμε έτσι καλύτερα τον δημιουργικό τομέα. Για παράδειγμα, να στηρίξουμε ίσως περισσότερο τις μη ε, κερδοσκοπικές επιχειρήσεις τις δημιουργικές, τα μουσεία, οικαστικές τέχνες κτλ. Επίσης, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, βεβαίως συμφωνώ με αυτά που μας είπατε, αλλά κατά τη γνώμη μου, η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας είναι και βεβαίως ε, και της Κομισιόν, της Νέας Κομισιόν, να προστατεύσουμε λοιπόν τα κονδύλια για την κουλτούρα, να μην θεωρούνται σαν κονδύλια οποιαδήποτε μέσα στον προϋπολογισμό. Η πολιτιστική ηθαγένεια είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρξει πολιτική ηθαγένεια. Και αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και σε επίπεδο προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ε, ερώτηση σας, δεν ξέρω σε ποιο έγγραφο της Επιτροπής το είδατε. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε φρασιολογία, χρησιμοποιούμε συνώνυμα, διαφορετικούς όρους, αλλά εμένα μου αρέσει η ιδέα της ε, δημιουργικής βιομηχανίας, του δημιουργικού κλάδου. Γιατί αυτό μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Ε, ζούμε σε ένα πολύ σύνθετο κόσμο και βεβαίω δημιουργία είναι πιο ωραίο όρο από το περιεχόμενο, αλλά είναι σχεδόν συνώνυμα πλέον. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνία και την καινοτομία, νομίζω ότι οι δράσει του Creative Europe πηγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στηρίζουμε ε, παραγωγή ντοκιμαντέρα, αλλά και φιλμ αρχείων και άλλες πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το παραμελούμε. Ναι, είναι βιομηχανία, είναι περιεχόμενο, αλλά είναι και ένα οικοσύστημα πολύ πιο ευρύ. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπατε, ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η Επιτροπή έκανε μια πρόταση για αύξηση λοιπόν του προπολογισμού, είναι η θέση της Επιτροπής και βεβαίως γίνονται διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό, όπως πάντα θα είναι πολύπλοκες. Ποια θα είναι η στρατηγική της επόμενης επιτροπής. Χρειαζόμαστε πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και για να διατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι λοιπόν μείζον το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. First of all, uh, Ο κύριος Κολάτζα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Βιόλα, που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστώ και για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Μιλήσατε για την AVMS Directive. Το άρθρο 23 στο εδάφιο Β λέει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν θα οδηγούν σε εξάντε έλεγχο η εφαρμογή κανόνων για το περιεχόμενο. Τι κάνει η Επιτροπή για να το διασφαλίσει ότι τα κρατη θα εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς σωστά. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και δεύτερο, για την ουδετερότητα του δικτύου. Η έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού για το Open Internet Access, για την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στα συμπεράσματα κατέληγε ότι δεν υπάρχει λόγος τροποποίησης της νομοθεσίας. Όμως η Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή και αναφέρει την υπόρξη πολλών προβλημάτων προσφορές με μηδενική αξιολόγηση, πλήρη απουσία διατάξεων πέναλτι κυρώσεων από κράτη-μέλη, το γεγονός ότι τα ε, μεγάλα μέσα ενημέρωσης το ε, κυριαρχούν επ' αυτού σε βάρος των μικρότερων. Θα τα δει όλα αυτά η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το πρώτο ερώτημα. Νομίζω ότι η οδηγία καταλήγει σε ένα πολύ λεπτό σημείο ισορροπίας που θα πρέπει κανείς να το διαβάζει ξανά και ξανά όταν σκοπό έχει να νομοθετήσει για θέματα παράνομου περιεχομένου στις πλατφόρμες ε, HVMS. Η οδηγία έχει ένα τρίγωνο. Έχουμε την αξιοπρέπεια στη μία γωνία, το παράνομο περιεχόμενο και ε, λόγος που μπορεί να πλήξει ε, διαφόρους και κυρίως τα παιδιά και τρίτο, ε, σε τρίτη γωνία είναι η ελευθερία του λόγου. Το σημαντικό δηλαδή είναι η ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών σημείων και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει εδώ μετά από 7 τριμερείς διαλόγους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λειτουργήσει πράγματι προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι η οδηγία το επιτυγχάνει, διότι αναφέρει ξεκάθαρα ότι πρέπει να τηρηθεί αυτή η συμφωνία δηλαδή. Ο καλύτερος τρόπος διατήρησης ισορροπίας είναι να έχουμε ένα σύστημα ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών οι οποίε θα είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Διότι ε, στη τελική οι αποφάσει θα λαμβάνονται αναπερίπτωση. Το σύστημα ε, ε, περιλαμβάνει μια προσέγγιση σε δύο βήματα. Πρώτον, στις γενικές ώρες οι πλατφόρμες πρέπει στους γενικούς όρους οι πλατφόρμες πρέπει να δηλώσουν ότι συμμορφούνται με αυτές τις αρχές της οδηγίας και το πράττουν. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό υπάγεται στην αυτορύθμιση, έστω. Αλλά δεν θα επηρεάσει τα, ε, το περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Μετά μπορεί κάποια ρυθμιστική αρχή να παρέμβει και να προσφύγει. Άρα θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση της ισορροπίας εκεί. Πώς ξέρουμε ότι η παρέμβασή μας θα είναι αντικειμενική. Διότι ο νομοθέτης, η ρυθμιστική αρχή, δεν θα επηρεάζεται από την κυβέρνηση. Δεν είναι αυτός που θα πει στον ε, ε, στη ρυθμιστική αρχή τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Η συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών θα εγγυηθεί ότι ε, το σύστημα θα διατηρήσει αυτή την ισορροπία μεταξύ αξιοπρέπειας, ελευθερίας λόγου και προστασίας. Όλα αυτά είναι η βάση της συμφωνίας. Είναι λεπτή η ισορροπία, αλλά ο μηχανισμός νομίζω έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να κατοχυρώνει, να εγγυάται αυτή την ισορροπία. Τώρα για την ιδιαιτερότητα του δικτύου. Ο σχετικός κανονισμός δεν είναι τέλειος, τίποτα δεν είναι τέλειο σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά είναι ο βέλτιστος δυνατός. Ε, σε όλο τον κόσμο οι καλύτερες διατάξεις είναι αυτές που έχουμε εμείς για την ουδετερότητα του διαδικτύου. έχει ένα αποτέλεσμα ήδη σημαντικό σε ό,τι αφορά την προστασία του πολίτη, των startup και το καθεξής. Γνωρίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το zero rating. Ε, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να σταματήσουν το zero rating σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους. όσοι θέλουν να ξανοίξει το κεφάλαιο για την ιδιαιτερότητα του δικτύου. Εάν το επιτύχουν αυτό θα είναι πιο κοστοβόρο, πιο διαπανηρό ή πιο ισορροπημένο. Θα καταλήξουμε με ένα καλύτερο προϊόν ή με ένα χειρότερο προϊόν. Τίθεται αυτό το ερώτημα. Εντύπωση μας είναι ότι σήμερα το καλύτερο που μπορεί κανείς να κάνει για να προστατεύσει τις αρχές του κανονισμού και για να διατηρήσει αυτή την ισορροπία μεταξύ της ε, ε, ε, ε, την ισορροπία μεταξύ όλων αυτών είναι να τα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να έχουμε τακτές εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και βεβαίως να αφήσουμε ενδεχόμενα να αλλάξουμε και άποψη του χρόνου. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω ότι επειδή η διορμηνία θα σταματήσει ακριβώς και μισή, θα ήθελα να μου πείτε ποιος ε, δεν μπορεί να μιλήσει αγγλικά, να κάνει την ερώτησή του στα αγγλικά. Ε, δείξτε κατανόηση. Θα δω, πάρουμε πρώτα την κυρία Καμερβέρτ και μετά οι υπόλοιποι στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φόντερ Λάιν στις 16 Ιουλίου συζήτησε το θέμα του Service Act όσον αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα προσφέρονται και θα διοχετεύονται και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι για μας αρκετά σαφές το γεγονός του πώς ακριβώς θα διασφαλιστεί εδώ η ελευθερία έκφρασης, μια βασική αρχή θα ήθελα να ακούσω κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο από εσά. Πώς το οραματίζεστε αυτό. Η ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ επίσης. Εμείς ε, ξέρουμε ότι όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων, στην πράξη ε, ε, το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ ικανοποιητικό και πολύ επιτυχές. Μπορεί η Επιτροπή να μας δώσει στις διάφορες χώρες, στα διάφορα κράτη-μέλη, μία λίγο πιο λεπτομερή αποτίμηση και απολογισμό του πώς υλοποιούνται όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό για τους νέους. Επίσης μας ενδιαφέρει τι μέτρα έχουν υλοποιηθεί από τα κρατημέλη. Το άρθρο 6 συγκεκριμένα του κανονισμού προϋποθέτει μία πολύ συγκεκριμένη φάση υλοποίησης. Τι κάνει η Επιτροπή, παρακολουθεί, ρωτάει, υπάρχουν μηχανισμοί κυρώσεων όσον αφορά την μη εφαρμογή, τη μη έγκαιρη εφαρμογή. Τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή έτσι ώστε να κινητοποιήσει λίγο τα κράτη-μέλη τα οποία δεν επιταχύνουν τις διαδικασίες. Ο κύριος Βιόλα θα απαντήσει σε ερωτήσεις από κοινού. Κυρία Μαντένη, έχει το λόγο. Κάντε την ερώτησή σας. Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου αφορά το blog σας. Το Φεβρουάριο μιλήσατε για το διαδίκτυο των ανθρώπων. Όλοι ακούσαμε ανησυχίες όσον αφορά την ψυχική υγεία, την πνευματική υγεία παιδιών και νέων, ανήλικων και νέων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, και η ερώτηση μου αφορά και τις πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς ε, διαπραγματεύεστε και με τους γίγαντες ε, του τομέα, του διαδικτύου και με τους εμπειρογνώμονες. Πέρα δηλαδή από το θέμα του κέρδους. Έχετε λάβει υπόψη σας όλες αυτές τις ανησυχίες για την πνευματική υγεία των νέων και των παιδιών και τη διασφάλισή τους. Έχω κάποια νέα παιδιά που θα έρθουν από την Αγγλία ε, στις Βρυξέλλες. Με μεγάλη χαρά θα σας καλούσα αν μπορείτε να έρθετε να τους συναντήσετε. Η τελευταία ερώτηση θα γίνει από μένα. Εγώ θα, μιλ... θα ήθελα να θίξω το θέμα του Euronews. Αύριο έχουμε εδώ την επεξεργασία της έκθεσης που αφορά το Euronews ε, από μέρους του ελεκτικού συνεδρίου. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω από σας από την Επιτροπή, όσον αφορά τα διάφορα σημεία που αναφέρει η έκθεση αυτή.